Bueno, pues buenas tardes. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Si les parece, comenzamos con el orden. Παρακαλώ, ας αρχίσουμε με, την ημερήσια διάταξη. Σημείο 1 πρώτα, έγκριση της διάταξης. De πριν όμως από την έγκριση. relación con la... Πριν από την έγκριση επαναλαμβάνω να σας επισημάνω δύο τροποποίησεις. Στο σημείο 9, πρωτόκολλο Ελίες με το Μαυρίκιο και το 13, έχουν αναβληθεί για την επόμενη συνεδρίαση. Οπότε τα σημεία 9 και 11 δεν πρόκειται να τα εξετάσουμε. Και τα σημεία 15 και 17 θα τα 15 ε, και 16 θα τα αντιστρέψουμε στη συζήτηση. Δηλαδή θα συζητήσουμε πρώτα το 16 και μετά το 15. Ξέρετε ότι δεν μου αρέσει καθόλου να τροποποιούμε την ημερήσια διάταξη. Αλλά με τις αλλαγές αυτές σήμερα θα έχουμε υπερφορτωμένη ημερήσια διάταξη, ενώ αύριο το πρωί θα έχουμε πολύ πιο ελαφριά ημερήσια διάταξη, μια και την απαλλάξαμε ήδη από δύο σημεία. Άλλε αλλαγέ όμω δεν μπορούμε να κάνουμε, γι' αυτό τι αφήνουμε έτσι. Σημείο λοιπόν 1. Έγκριση τη τροποποιημένη ημερήσια διάταξη. Σημείο 2. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων 28 και 29 Νοεμβρίου και 17-18 Δεκεμβρίου. Όπω πάντα, αν δεν υποβληθούν αντιρρήσεις ε, ή ενστάσεις μέχρι το τέλος ε, της σημερινής μας συνεδρίασης θα θεωρηθούν ως συγκεκριμένα. Σημείο 3. Ανακοινώσει του Προέδρου. Έχω μια ανακοίνωση, έναν αποχαιρετισμό. Ο Κλώδιο Καρέντα από τη Γραμματεία μας ε, ανακοίνωσε σήμερα και επίσημα ότι θα αλλάξει τον αέρα του. Αφήνει την αλία Γι' αυτό και τον αποχαιρετούμε επίσημα και τελετουργικά σήμερα, ευχαριστώντας το θερμά για τη συμβολή του σε όλο το διάστημα που συνεργάστηκε μαζί μας. Όχι μόνο κατά τη διάρκεια της δικής μου προεδρίας, αλλά και προηγουμένως. Θα ήθελα λοιπόν να το ευχηθώ καλή τύχη στα νέα του καθήκοντα και είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα είναι εξίσου αποτελεσματικός και επιτυχημένος και στα καθήκοντα όπως είδα και στην Αλία. Αυτά λοιπόν και καλή σας τύχη. Περνάμε τώρα στο σημείο 4 της ημερής σας διάταξης. Το πρωτόκολλο δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας σχετικά με το καθορισμό των ελευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη Συμφωνία Αλληλευτικής Σύμπραξης μεταξύ των δύο πλευρών. Όπως ξέρετε, ήδη για το θέμα αυτό έγινε κάποια ανταλλαγή απόψεων και σε μια συνεδρίση των συντονιστών ανέκυψε η πιθανότητα να προσκαλέσουμε ένα μικρό αριθμό εμπειρογνωμόνων και τους ευχαριστώ θερμά που ανταποκρίθηκαν στην τελευταία στιγμή πρόσκληση γιατί θα μας παρουσιάσουν τις απόψεις τους για το θέμα αυτό. Είχαμε καταρχήν πέντε εμπειρογνώμονες που ορίστηκαν από τις πολιτικές ομάδες για να μας διαφωτίσουν σήμερα. Το Δοχον Κάρλος Μαρτίν Φραγκέιρο που τελευταία στιγμή ανακοίνωσε ότι κολλείεται. Οπότε από τους πέντε μας έμειναν τέσσερις καλεσμένοι, τέσσερις εμπειρογνώμονες. Εγώ θα έλεγα να διαχωρίσουμε σε δύο τμήματα την ακρόαση αυτή. Στο πρώτο τμήμα να ακούσουμε τους εμπειρογνώμονες και να ακολουθήσει μια ανταλλαγή απόψεων των μελών της Επιτροπής με τους εμπειρογνώμονές μας, να υποβληθούν απορίες, ερωτήσεις, να διαλευκαθούν κάποια θέματα και αφού ολοκληρώσουμε αυτή την πρώτη ενότητα με την ακρόαση των εμπειρογνωμόνων και τη συζήτηση στην Επιτροπή, να περάσουμε στην δεύτερη ενότητα που, όπου θα παρουσιαστεί η γνωμοδότηση από τον υποφαινόμενο με συζήτηση βέβαια μετά. Πρώτος γύρος λοιπόν ακρόαση των εμπειρογνωμόνων και συζήτηση μαζί τους και δεύτερη ενότητα παρουσίαση της έκθεσης από τον πρόεδρο, τον εισηγητή και μετά συζήτηση. 10-12 λεπτά στον καθένα θα δώσουμε, το πολύ 15, αλλά παρακαλώ να μην τα ξεπεράσετε τα 15 λεπτά, μια και από 5 γίνατε 4 και μετά την παρουσίαση του κάθε εμπειρογνώμονα. Θα παρακαλούσα τον επόμενο εμπειρογνώμονα να μην επαναλαμβάνει σημεία που έθιξε ο προηγούμενος ομιλητής για να μην έχουμε επικαλύψεις και επαναλήψεις και να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το χρόνο μας. Χωρίς άλλη λοιπόν καθυστέρηση θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Μπενουά Καγιάκ που είναι διευθυντής μελετών στο Ινστιτούτο Οκεανογραφικών Εξελίξεων. Του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Θα σας παρουσιάσω κάποια στοιχεία όσον αφορά την εκμετάλλευση των αποθεμάτων στη Μαυριτανία έχοντας αναλύσει το θέμα εις βάθος και έχοντας προβεί σε αξιολόγηση της συμφωνίας, του πρωτοκόλου συμφωνίας που εξέπνωσε το 2012. Θα σας παρουσιάσω κάποια στοιχεία όσον αφορά τα αποθέματα ε, του χταποδιού. Να σας δώσω κάποια στοιχεία. Στη Μαυριτανία η επίσημη αξιολόγηση των αποθεμάτων των ε, χταποδιών γίνεται κάθε τετραετία στα πλαίσια εργασιών από το Εθνικό Ινστιτούτο Ερευνών και πιο συχνά στα πλαίσια του ΚΟΠΑΣ που είναι ο φορέας του ΦΑΟ που ε, δίνει επιστημονικές συμβουλές. Τελευταίες γνωστές αξιολογήσεις και στοιχεία που έχουμε ε, αφορούν έρευνα που έγινε το 2009 στην ΚΟΠΑΣ και το 2010 στην Επιστημονική ε, Επιτροπή του ΜΟΠ. Αξιολόγηση του 2009 συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία μέχρι το 2008 και αξιολόγηση του 2010 τα στοιχεία μέχρι το 2009. Μέχρι το 2009 Ξέρουμε ότι η Αλία έδειχνε δείκτες στο ερυθρό, στο κόκκινο, διότι η βιομάζα των χταποδιών ήταν 85% της ε, βιομάζας ε, που ήταν σε ισορροπία, NSY, και η ελευτική προσπάθεια ήταν υπερβολική, διότι στα 155% της επιτρεπόμενης αληφτικής. Οι γνωματεύσεις των εμπειρογνωμόνων έκαναν την ίδια σύσταση. Η προσπάθεια όσον αφορά το χταπόδι έπρεπε να μειωθεί. Αυτό ήταν το 2010 η αποτίμηση. Μετά την αξιολόγηση της ομάδας εργασίας του 2010, από ό,τι ξέρουμε έκτοτε δεν έγινε αξιολόγηση, είναι ένα κάτι που πρέπει να ξαναγίνει. Όμως, το Επιστημονικό Ινστιτούτο της Μαυριτανίας, το IMROP, παρακολουθεί το απόθεμα χτωπαδιών ε, και μηνύα προσπαθεί να κάνει την αποτίμηση στις θάλασσες. Τα γραφήματα που βλέπετε δείχνουν τα αποτελέσματα, τους δείκτες αυθονίας που ε, συνελέχθησαν από τη θάλασσα. Δεν ξέρουμε καλά, δεν βλέπουμε καλά την κλίμακα του ιστογράμματος αυτού, αλλά η δεξιά κολόνα αφορά τον Ιούλιο του 2012 και ξεκινάει το ιστορικό το 2008 των στοιχείων. Αυτό που βλέπουμε το 2012 είναι ότι οι δείκτες είναι αρκετά ψηλοί, σχετικά ψηλοί, που φαίνεται να δείχνουν μια καλύτερη κατάσταση όσον αφορά τους σπόρους και πρέπει να επιβεβαιωθεί η τάση αυτή, έτσι δεν περαιτέρω, διότι μετά τις μετρήσεις του Ιουλίου 2012 η όλη μορφή της αλληλείας άλλαξε με την πάυση των αλλιεύσεως των ευρωπαϊκών κεφαλόποδων. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Έχουμε παλιά στοιχεία που δεν είναι ακόμα επισημοποιημένα. Χρειάζεται νέα αξιολόγηση των αποθεμάτων χταποδιού, επίσημη αποτίμηση και η τιμή του MSY. Διότι ήταν 30.000 τόνους εκτίμηση επί μακρόν. Ο τρόπος όμως της αλληλείας όσο αλλάζει και άλλαξε διότι τα ευρωπαϊκά σκάφη σταμάτησαν την αλληλεία και είδαμε σημαντική αύξηση της αλίας σε επίπεδο ε, ε, βιοτεχνικό. Και ίσως να έχει αλλάξει η τιμή του MSY. Αλλά χρειάζεται μια νέα αξιολόγηση του αποθέματος για να δούμε τι γίνεται, ποια είναι η σχέση αλίας με την ισορροπία. Εάν ε, πρέπει να γίνει κάτι ή όχι, αν τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Αυτά για το χταπόδι. Για τα μικρά πελαγικά είδη στη Μαυριτανία αυτή η αλία ε, αφορά τα ψάρια που κατανοούνται επί τόπου. Υπάρχει αρκετή αυθονία εδώ και δεκάδες χρόνια. Υπήρξε και βιομηχανική εκμετάλλευση από μεγάλα λευτικά ευρωπαϊκά, ρωσικά, ουκρανικά Εδώ και δύο χρόνια περίπου αυξήθηκε το ενδιαφέρον για τα μικρά πελαγικά είδη, διότι αυξήθηκε η παγκόσμια τιμή των ηχθιαλεύρων. Η αύξηση της τιμής οδήγησε στο να διαφερθούν οι αλείς και στα ανατολικά του ειρηνικού αυξήθηκε η ζήτηση και στη Μαυριτανία κατασκευάστηκαν εργοστάσια αλεύρων. Και κινεζικέ πολυεθνικέ, ο όμιλος κινέζικος, ετοιμάζει να κάνει αρκετά μεγάλες επενδύσεις στον τομέα αυτό για την παραγωγή χθιαλεύρων στη Μαυριτανία. Νοπάψα χρησιμοποιούνται για τα αλεύρα, τροφοδοτούνται τα εργοστάσια από, από τη Σενεγάλη, από βιοτεχνική αλία της Σενεγάλης με νοπά ψάρια και από τοπικά μικρά ψαράδικα σκάφη. Στα σαρδελοειδή είναι άγνωστη, σαρδελόρεγγες είναι άγνωστη η κατάσταση. Η Κόπας έκανε μία αποτίμηση το 2010 και συνεπέρανε ότι από θέματα στις σαρδελόρεγγες ε, θεωρείται ότι υπεραλλιεύονται. η ΚΟΠΑΣ αμφισβητεί την ορθότητα της αξιολογήσεως, διότι εδράζεται επί στοιχείων ε, που δεν καλύπτουν ε, πλήρως τους στόλους που αλλιεύουν. Η διάγνωση οδηγεί στην ε, υπερεκμετάλλευση, αλλά τα στοιχεία δεν είναι πάρα πολύ βάσιμα αξιο, αξιόπιστα, χρειάζεται μια άλλη αξιολόγηση των αποθεμάτων. Να υπογραμμίσουμε ότι οι σαδελόρεγγες ανήκουν στα μικρά πελαγικά είδη, αφορούν Νότια Σενεγάλη, Μαρόκο, τις παράκτιες χώρες και δεν υπάρχει διεθνή συμφωνία της διαχείρισης αυτών μεταξύ αυτών των χωρών της Δυτικής Αφρικής όπως η σύμβαση του ΟΗΕ για, τα, για το δίκαιο της θαλάσσης θα απαιτούσε. Τα μικρά αυτά πελαγικά είδη ε, δεν έχουν προσαρμοστεί δεόντως στις ε, σημερινές ανάγκες όσον αφορά τη διατήρηση των αποθεμάτων. Να πω, να πω μερικά πράγματα όσον αφορά το πρωτόκολλο της συμφωνίας που διαπραγματευτήκαμε εδώ και μερικούς μήνες. 1η Αυγούστου του 2012 τέθησε ισχύ. σημείο τα γεγονότα πέρα από τη μείωση του δυναμικού αλίευσης που σταμάτησαν οι ευρωπαϊκές, τα ευρωπαϊκά αλλιευτικά την αλίευση κεφαλοπόδων λόγω εξάρτησης αποθεμάτων ε, και υπάρχει ο περιορισμός ζωνών στα ανοιχτά, αλλιευτικών ζωνών. Για τις αδελόρεγγες απομάκρυνση από τις ακτές είναι να μειωθεί η πίεση στις υπερεκμεταλλευόμενες ε, στα υπερεκμεταλλευόμενα είδη και να ενισχύσουμε τις, ε, τους ντόπιου ε, μικρούς στόλους, τεχνικούς στόλους. Η κυβέρνηση της Βρετανίας στηρίζει την βιοτεχνική αλία και δίνει περισσότερο χώρο σε αυτά τα σκάφη. Οι Σαδελόρεγγες σαν πηγή είναι μεταβλητή στον Ευρωπαϊκό Αλληλευτικό Στόλο. Έχουμε παράκτια πηγή, πόρο, ε, και στα πιο ανοιχτά. Εστονία, Λιθουανία αλλιεύουν κάποια είδη ε, που είναι, ανήκουν στα μικρά ε, πελαγικά αλλά δεν ανήκουν στις αρδελόρεγγες. Λοιπόν, οι ζώνες προωθη... αλίας προωθήθηκαν προς τα ανοιχτά για να προστατευτεί και η βιοτεχνική αλία και να μειωθεί ο αρνητικό αντίκτυπος στο περιβάλλον. Διότι παράκτη αλία γίνεται σε βάθος μέχρι 20 μέτρα περίπου. Στα ανοιχτά πάει μέχρι 100 μέτρα Και όσον αφορά και την παραλίευση ε, υπήρχαν αρνητικές συνέπειες όσον αφορά την αλία την παράκτεια. Μεγαλύτερη, μεγαλύτερο αντίκτυπο είχε. Όσον αφορά τις άδειε τώρα, από το προηγούμενο πρωτόκολλο άλλαξαν τα πράγματα. Η τιμή της άδεια επανεξετάστηκε, αναθεωρήθηκε, άλλαξε και ο τρόπος υπολογισμού και ο τρόπος ισχύω βασίζεται με το βάρος, με τους τόνους. σχέση τιμής που πληρώνουν οι ναυλωτές για την πρόσβαση σε σχέση με τη μέση τιμή που μπορούμε να ελπίζουμε μέσω της αλίευσης. Για τα σκάφη αλίας γαρίδας 7.500 ευρώ ένα τόνο πληρώνεται για τις γαρίδες. 6.020 ένα τόνο. Ε, σχέση, ε, είναι η άδεια. 8% σχέση. Η άλλα είδη 1500 ευρώ το τόνο, η εισφορά είναι 300 περίπου ευρώ τον τόνο, μια σχέση 2%. Για τα μικρά πελαγικά, αν πάρετε βάση τιμή του αλλιεύματος 600 τόνο είναι πιο φτηνά τα μικρά πελαγικά είδη από τα άλλα είδη. Η εισφορά 123 ευρώ τόνο σχέση 20%. Αυτά τα στοιχεία σας δείχνουν ότι υπάρχουν διαφορές, αρκετές διαφορές μεταξύ των κατηγοριών. Μεταξύ αυτού που πληρώνουν οι ναυλωτές για την πρόσβαση και των τιμών που μπορούν να πετύχουν μέσω των αλευμάτων τους. Ε, αυτά είναι κάποια στοιχεία τα οποία θα να σας παραθέσω και ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Καγιάρ για την ε, παρουσίαση. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Γκέρτ Βαν που είναι πρόεδρος της ε, Ένωσης ε, Διοκτητών ε, Μηχανότρατων Ψυγείων για την Πελαγική Ελία. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που με καλέσατε σήμερα εδώ στη σημερινή συνεδρίαση. Είμαι ο πρόεδρος αυτής της ε, Ένωσης ε, για τα πελαγικά ψυγεία, για τις μηχανότρατες ψυγεία. Εκπροσωπούμε αρκετές ενώσεις στην Δυτική Αφρική. Θα ήθελα να σας δώσω κάποια στοιχεία για το πώς ε, βλέπουμε εμείς την ε, κατάσταση αυτή με την συμφωνία την αλληλευτική με τη Μαυριτανία. Για τον, την πελαγική πτυχή του θέματος. Καταρχάς, το σημείο εκκίνησης ως τομέας ποιο ήταν αυτό, το σημείο εκκίνησης που είχαμε. Εμείς ήμασταν πάντα υπέρ ε, της σύναψης τέτοιων συμφωνιών με τη Μαυριτανία. Πολλές φορές είπαμε ότι μπορεί να προτιμούμε μια ιδιωτική συμφωνία, αλλά πάντοτε υποστηρίζαμε Τέτοιε αλλιευτικέ συμφωνίε μεταξύ ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και Μαυρετανία. Επίση, πάντα, και ακόμα την έχουμε, η θέση μα ήταν ότι θα πρέπει να υπάρξει ε, συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα κράτη-μέλη, τι κυβερνήσει του για όλα τα θέματα που αφορούν την αλληλεία. Όχι μόνο για την εξωτερική διάσταση, αλλά για ό,τι άπτεται τη πολιτική αλληλεία. Επίση, έχουμε ενεργή δράση στην Μαυρετανία από το 1995, περίπου 17-18 χρόνια τώρα, ξεκινήσαμε με μια ιδιωτική συμφωνία. Τότε δεν υπήρχε βεβαίω η απαλλαγική πτυχή στην Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Βρετανία και αμέσω μετά η Κομισιόν μα κάλεσε να ενσωματώσουμε αυτή την ιδιωτική συμφωνία σε μια Ευρωπαϊκή Συμφωνία με την ε, Μαυρετανία και το οποίο συμφωνήσαμε. Και από τότε αλλιεύουμε στα πλαίσια τη Συμφωνία τη Ευρωπαϊκή. Γενικώ, Τώρα ε, θεωρούμε ότι είναι καλύτερο να, έχουμε, να μην υπάρχει συμφωνία από το να υπάρχει μια κακή συμφωνία. Και αυτό είναι ένα συμπέρασμα στο οποίο θα καταλήξω κατά τη διάρκεια της ε, παρουσίασης ότι η, αυτή η τρέχουσα συμφωνία είναι κακή συμφωνία σε ό,τι αφορά τα πελαγικά είδη. Να σας πω τώρα εδώ κάποια στοιχεία για να συγκρίνετε σε σχέση με την ε, παλαιά συμφωνία για το απόθεμα. Οι ε, ευκαιρίε αλλήλευση ε, ε, ήταν 300.000 τόνοι το χρόνο. Δεν υπάρχει εδώ πέρα διαφορά μεταξύ των δύο συμφωνιών. Έχει υπάρξει μια μικρή αύξηση του πληρώματο των Μαυριτανών. 60% ήταν, ενώ η παλαιά συμφωνία ήταν στο 37% των Μαυριτανών, που σημαίνει ότι έχουμε μια μικρή αύξηση του πληρώματος. Επίσης, τώρα ένα καινούργιο στοιχείο είναι ότι πρέπει να δώσουμε ένα, ε, δωρεάν ένα 2% των αλλιευμάτων ανα, ανα έξοδο για αλίευση. Ε, τέλος πάντων, ε, πιεστήκαμε λίγο για να γίνει αυτό. Ε, γιατί πολλέ φορέ χρειάζεται να δώσουμε αρκετού τόνου δωρεάν αλλιευμάτων και αυτό είναι ένα νέο στοιχείο σε τούτη την συμφωνία. 2% λοιπόν των αλλιευμάτων μα δίνεται δωρεάν. Επίση, έχουμε ένα ανώτατο όριο 2% περιθώριο ανοχής ανάμεσα στο μητρό, στις καταχωρήσεις στο μητρό και στις εκφορτώσεις. Η ευρωπαϊκή πελαγική ε, βιομηχανία δίνει ένα 10% επίπεδο ανοχής. Το 2% δηλαδή είναι πολύ περιθωριακό ακόμα και ως περιθώριο ανοχής. Δίνει δηλαδή τη δυνατότητα δεν θέλω να είμαι κοινικός, αλλά δίνει την ε, ε, δυνατότητα στους ε, πλειοκτήτες να έχουν μεγάλη διαφορά μεταξύ του εκφορτωθέντος αλλιεύματος και του ζυγισμένου αλλιεύματος. Και έτσι μπορούν να γλιτώσουν πολύ μεγάλα πρόστιμα. Τώρα έχουμε διπλό σύστημα δορυφορικό που ήταν υποχρεωτικό στην συμφωνία την καινούργια Έχουμε την ε, ε, υποχρέωση να μεταφέρουμε αλλιεύματα. Δεν υπήρχε ε, τέτοια υποχρέωση στην παλιά συμφωνία και επίσης υπάρχει μια εξαίρεση για κάποια σκάφη τα οποία δεν μπορούν να κάνουν αυτή την μεταφορά, την μεταφόρτωση. Εδώ τώρα είναι η μεγάλη διαφορά που υπάρχει για το τέλος για τους πλειοκτήτες. Στην παλιά συμφωνία πληρώναμε περίπου για ένα μεσαίο σκάφος 50.000 ευρώ το μήνα και αυτό έχει αυξηθεί δραματικά και φτάνει περίπου τους 300, τα 300.000 ευρώ τον, το μήνα για ένα πάλι μέσο σκάφος. Ε, Βεβαίω αυτό θα μπορούσατε να το δείτε και αν συγκρίνετε και τις ε, υπόλοιπες κατηγορίες ανάμεσα στην παλιά και την νέα συμφωνία. Πληρώνουμε πολύ περισσότερο τώρα και για τις υπόλοιπες ε, κατηγορίες. Και το τελευταίο είναι το αλληλευτικό όριο. Έχουν υποθεί πολλά για το αλληλευτικό όριο. Έχει γίνει όριο, ε, το, έχουν γίνει όριο τα 20 μίλια, τα 20 ναυτικά μίλια. Στην παλαιά συμφωνία ήταν 12 με 13 τα μίλια, ανάλογα με την ε, συμφωνία. Ε, από το 1995 ήταν έτσι η κατάσταση. Πάντα ήμασταν στα 12-13 μίλια και τώρα είμαστε στα 20. Έχει αυξηθεί λοιπόν αρκετά και μάλιστα εν μία νυχτή. Να μπω λίγο σε κάποιες λεπτομέρειες για αυτό το όριο, την αλλαγή που έγινε. Προτάθηκε από την Μαυριτανία, από την διαπραγματευτική ομάδα το Δεκέμβρη του 2011. Οι λόγοι για τους οποίους προτάθηκε δεν ήταν απόλυτα σαφείς. Ε, θα μπορούσε κανείς να πει ότι ήθελαν να προστατεύσουν ε, την ε, φρίσα ε, αλλά πάλι δεν ήταν και σίγουρο ότι αυτό ήταν ο λόγο. Επίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κρατημέλη αποφάσισαν ότι θα αποδεχτούν αυτό τον λόγο, παρά το ότι εμεί, η βιομηχανία δηλαδή, ο κλάδο, ήθελε, ήθελε το αντίθετο. Επίση, από την αρχή είχαμε πει ότι ε, αυτό ήταν λόγο για να μην υπάρξει συμφωνία. Ήμασταν απόλυτα σαφεί και στα κρατημέλη και στην Κομισιόν ότι αυτό θα σημαίνει ουσιαστικά ε, μη επικερδή αλληλεία και αυτόματα θα οδηγούσε σε πολύ χαμηλή, ίσως και μηδενική χρήση του, της πελαγικής πτυχής της αλίας. Οι τελευταίες διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν Ε, Βεβαίω, ε, πάντα ε, στι τελευταίε διαπραγματεύσει ε, παρεμβαίναμε εμεί με επιστολέ μα, με παρεμβάσει μα. Η Κομισιόν ζήτησε από τα κρατημέλη να, να τι δώσουν κάποια αριθμητικά στοιχεία για την αλληλευτική του θέση για το 2011. Αυτό δόθηκε από τα κράτη-μέλη στην Κομισιόν πριν τον τελευταίο γύρο των διαπραγματεύσεων που ήταν τον Ιούλιο του 2012 και να σας ε, πω κάποια πράγματα για τα δικά μας τουλάχιστον τα σκάφη. Για την Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις κάτω χώρες που ε, είναι ενεργά στην ε, Μαυριτανία. Καταρχάς έχουμε τον, το όνομα του σκάφους, μετά έχουμε το ποσοστό αλλιευμάτων του 2011 που έχουν γίνει εντός των, των ναυτικών ορίων, δηλαδή εντός των 13 έως 20 ναυτικών μιλίων και η τρίτη στήλη είναι τα αλλιεύματα του 2011 που είναι εκτός του ορίου των, ναυτικών, των 20 ναυτικών μιλίων. Κατά μέσο όρο ο στόλος μας, βλέπετε και τα ονόματα των σκαφών από κάτω, κατά μέσο όρο το 2011 ο στόλος μας, PFA, ε, αλίευσε 56% των αλλιευμάτων εντός των ορίων των 20 μιλίων και 44% εκτός αυτών. Αν δείτε τα ποσοστά θα δείτε ότι υπάρχει βεβαίως και διαφορά ένα σκάφος. Τα περισσότερα σκάφη δεν, είναι, ε, δεν ήταν ενεργά καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, κάποια ήταν. Κάποια ε, ήθελαν να αλλιεύσουν κατά τη διάρκεια της ε, ε, περίοδου σαρδέλ, αλλιεύσης σαρδέλας που είναι εκτός των 20 ναυτικών μιλίων αλλά παρόλα αυτά μπορείτε να δείτε γενικώ ότι υπάρχει μεγάλη εξάρτηση της αλληλείας εντός των 20 ναυτικών μιλίων, εντός αυτού του ορίου. Αν δείτε τώρα τον πολωνικό στόλο, Έχουμε δύο εδώ σκάφη. Δεν έχω ε, τα στοιχεία για τη Λιθωνία και τη Λετωνία, αλλά η Πολωνία που μου έδωσε τα στοιχεία, τα έχει και η Κομισιόν βεβαίω αυτά, βλέπετε ότι δύο ε, πολωνικά σκάφη ε, εξαρτώνται ακόμη περισσότερο από την ελίευση εντό των 20 ναυτικών μίλιων. Ο πολωνικό στόλο κυρίω ασχολείται με την αλίευση σαφριδιού και λιγότερο φρύσα. Αλλά εμεί αλλιεύουμε το αντίθετο και το σαφρίδι, ε, για το σαφρίδι η, ε, ε, εξάρτηση εντός των 20 μιλίων ήταν πολύ μεγαλύτερη από τη δική μας. Τώρα, κάποια συμπεράσματα για την, για την πελαγική οπτική και κλείνω. Σας έδωσα κάποιες τεχνικές τις συνθήκες ε, το βασικό είναι ότι υπάρχει ε, δραματική αύξηση της, ε, του τέλους άδειας, το οποίο έχει οδηγήσει σε, πολύ λιγότερη χρήση της, του πρωτοκόλου που έχει συμφωνηθεί για την παλαιγική αλλιεύση που σημαίνει ότι υπάρχουν λιγότερα αλλιεύματα επομένως δεν υπάρχει κέρδος από τότε τη συμφωνία. Μετά, η επέκταση του αλληλευτικού ορίου στα 20 ναυτικά μίλια είναι πραγματικά αυτό που θα έπρεπε να ακυρώσει την όλη συμφωνία. Επίσης, σε κάθε επίπεδο στην ε, Κομισιόν, αλλά και κάθε φορά που ε, γινόντουσαν διαπραγματεύσεις και σε κάθε γύρο διαπραγματεύσεων, λέγαμε ότι χωρίς αυτό το, 20, το όριο των 20 ναυτικών μιλιών θα μπορούσαμε να σκεφτούμε να υπάρχει ένα υψηλότερο τέλος για την άδεια. Ακόμα και με αυτές τις τεχνικές ε, συνθήκες. Αλλά ε, τώρα δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Γιατί σίγουρα αν πάμε στην Μαυρετανία με τέτοιες προϋποθέσεις δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε λεφτά, θα χάσουμε μάλιστα λεφτά. Οι ε, τράτες είναι όντως ε, δύσκολο είδος να, για τη διαχείριση. Έχουμε και αυτή την ε, επιβολή του 20, των 20 ναυτικών μιλίων, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολη η κατάσταση. Μετά, οι προτεραιότητες του ευρωπαϊκού στόλου, που σημαίνει ότι όλες οι συνθήκες που έχουν τεθεί για τον Ευρωπαϊκό Στόλο θα πρέπει να πληρούνται και από τη Μαυριτανία. Ακόμα και για συμφωνίες που έχει η Μαυριτανία με μη ευρωπαϊκούς στόλους. Αλλά και ο ευρωπαϊκός στόλος και οι διεθνείς στόλοι έχουν φύγει από την περιοχή αυτή από τον Αύγουστο. Οπότε το πλεονέκτημα αυτό της, ε, της προτεραιότητας ουσιαστικά μόνο επί χάρτου ισχύει. Δεν είναι πρακτικό ε, πλεονέκτημα για κανέναν. Επίσης θεωρούμε ότι αν εμείς ως ε, ευρωπαϊκός πελαγικός ε, εξακολουθήσουμε να είμαστε απόντες από τη Μαυριτανία, ε, προφανώς αυτό δεν βοηθά καθόλου το να υπάρξει σωστή αποτελεσματική διαχείριση της αλληλείας, τουλάχιστον για τα πελαγικά είδη. Και αυτό το χρειαζόμαστε. Το χρειαζόμασταν από την αρχή. Πάντα επενδύαμε χρήματα, επενδύαμε ε, χρόνο σε αυτή τη διαδικασία. Αν ξέρουμε τώρα ότι ο Ευρωπαϊκός τόλο δεν πρόκειται να να είναι παρόν στην Μαυρετανία, δεν, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε αποτελεσματικά την αλληλεία μας. Επίσης, τα περισσότερα αλληλεύματα από τη Μαυριτανία εξάγονται σε χώρες Δυτικής Αφρικής, από την, ε, από Ιγυρία, ε, το Μαλί, την Μπουρκίνα Φάσο, την Κάνα. Και εδώ υπάρχει μεγάλο κενό στην προμήθεια αυτών των, την τροφοδοσία αυτών των αγορών πια. Και αρχίζουν ε, εκεί να υπάρχουν προβλήματα γιατί ε, υπήρχε πολύ μεγάλη παραγωγή πελαγικών ειδών στη Μαυριτανία που τώρα δεν υπάρχει. Και δεν φτάνουν λοιπόν τα λιεύματα στις αγορές της Δυτικής Αφρικής. Θεωρούμε λοιπόν ότι η θέση μας είναι αυτή που ήταν πάντα. Εμείς ως κλάδος εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε μια τέτοια συμφωνία λευτικής σύμπραξης με τη Μαυριτανία, αλλά θα πρέπει να είναι και οικονομικώς βιώσιμη θα πρέπει να είναι αποτελεσματική, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τους τοπικούς αλληλείς. Ε, αλλά θα πρέπει να είναι και επικερδής για τον ευρωπαϊκό στόλο. Προς το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι ε, τίποτα από όλα αυτά η, η τρέχουσα συμφωνία. Οπότε θα πρέπει να τροποποιηθεί το υπάρχον πρωτόκολλο. Ελπίζουμε ότι και εσείς θα μπορέσετε να κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας για να πείσετε και την Κομισιόν και το ε, Συμβούλιο να συμφωνήσουν ότι πρέπει να τροποποιηθεί αυτό το πρωτόκολλο. Ευχαριστώ. Muchas gracias. Σας ευχαριστούμε, κύριε Βαμπάλσφορτ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος ε, Σινταμέντα Βέτ, που είναι πρόεδρος ε, της ε, Εθνικής Ομοσπονδίας Παράκτειας Αιλίας Μικρής Κλιμάκος Μαυριτανίας. Ευχαριστώ. Κύριε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ, κύριε Ισηγητά, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που δίνετε σε έναν ψαρά παράκτης αλίας της Μαυριτανίας να λάβει το λόγο στην Επιτροπή σας. Ονομάζομαι Σενταχμέντ Αμπέτ και είμαι πρόεδρος της οργάνωσης παράκτης αλίας μικρής κλίμακος της Μαυριτανίας. Όπως ξέρετε η Μαυριτανία είναι αναπτυσσόμενη χώρα. Πριν από 35 χρόνια η παράκτη αλία της Μαυριτανίας περιοριζόταν σε παραδοσιακές κοινότητες, του Σιμραγκουέν και του Σουαλόφ της περιοχής του Ντιάγκο. Αλλά η δραστηριότητα που αναπτύχθηκε τότε και συνέβαλε στο να γίνει η παράκτη αλία μοχλός οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας μας είναι η αλία του χταποδιού. Και μπορώ να σας μιλήσω γι' αυτό γιατί είμαι ο πρώτος που ασχολήθηκε με την αλία αυτή το 1978, με την αλία του χταποδιού. Τότε μάλιστα θυμάμαι ότι είμαστε μόνο 17 σκάφη παράκτιας αλίας. Μάλιστα ψαρεύαμε και άλλα ψάρια και σκυλόψερα μεταξύ των άλλων. Τόγιο το λέμε στα μαυριτανικά. Τα πουλούσαμε όμως τα ψάρια αυτά μόνο 7, ε, ουάγιας, δηλαδή 2 λεπτά το ευρώ το κιλό. Το 1978 λοιπόν ε, η Ιαπωνέζικη ε, Συνομοσπονδία, συνεταιρισμός, ε, ε μου έκανε ένα διάβημα και μου είπε ότι μπορούμε να αλλιεύουμε πολύ καλύτερης ποιότητας χταπόδι με δοχεία και μάλιστα θα παίρναμε και πολύ καλύτερες τιμές. Ξεκίνησε λοιπόν αυτή την αλία αχταποδιού με δοχεία. Μάλιστα έκανα δοκιμές με πολλά υλικά για τα δοχεία αυτή, με τσιμέντο, με πλαστικό, με ε, αλλά κανένα υλικό δεν ήταν ιδανικό για τη δημιουργία αυτών των δοχείων. Είτε ήταν πολύ έφραστα και έσπαζαν, είτε ήταν πολύ ελαφριά, είτε παρά ήταν βαριά. Πήγα όμω μια μέρα στη Λαπάλμα και διαπίστωσα ότι εκεί πουλούσαν νερό Ισπανί σε μπουκάλια 5 λίτρων, που ήταν ιδανικέ διαστάσει για τα δοχεία που έψαχνα εγώ για, το... για την αλία του χταποδιού. Πήγα λοιπόν ε, στον παρασκευαστή αυτών των ε, δοχείων νερού ε, παρήγγειλα πολλά και τα έστειλα στη Μαυριτανία. Το αποτέλεσμα ήταν καταπληκτικό για την αλία με τα μπουκάλια του νερού ουσιαστικά. Και μάλιστα μια και αυτό έγινε μετά την μεγάλη ξηρασία του 1973, πολλοί Μαυριτανοί μετατοπίστηκαν προς τις ακτές και άρχισαν να δουλεύουν αλλιεύοντας χταπόδι όπως εγώ δημιουργήθηκε και η εταιρεία της Μαυριτανίας για την εμπορευματοποίηση αλληλευτικών προϊόντων το 1984 για να προωθήσει τα προϊόντα αυτά. Σήμερα είμαστε 36.000 ε, ε, αλίες, παράκτες αλίες, με 7.500 σκάφη βιοτεχνικά και σε ό,τι αφορά την αλία του χταποδιού εξασφαλίζουμε 60% της εθνικής παραγωγής σε ποσότητα και 70% σε αξία. Μάλιστα δημιουργούμε το 90% των θέσεων απασχόλησης στον τομέα της αλίας. Μάλιστα με ε, κόσμο που εργάζεται σε 50 εργοστάσια ε, μεταποίησης ε, ή κατάψυξης, σε 12 εργα... εργαστήρια κατασκευής πυρογών, εκατοντάδες παρασκευαστές υλικού, μεταφορείς, κατασκευαστές δοχείων κτλ. Αυτά που σας διηγούμε λοιπόν εδώ είναι αυτό που εμείς αποκαλούμε ανάπτυξη στη Μαυριτανία. Βέβαια θέλουμε ταυτόχρονα να εντάξουμε την ανάπτυξη αυτή σε μια προοπτική αηφόρου βιώσιμη αλίας. Θα πρέπει λοιπόν να σας υπενθυμίσω ότι η αλία με το δοχείο είναι επιλεκτική αλία. Πιάνουμε λοιπόν το, το χταπόδι που κρύβεται στο βάθος του δοχείου και αν είναι πολύ μικρό αυτό το χταπόδι το επιστρέφουμε ζωντανό στη θάλασσα. Εμείς έχουμε στόχο να αλλιεύσουμε χταπόδι πρώτης ποιότητας. Γι' αυτό μικρά, τα μικρά χταποδάκια δεν είναι για μας από εμπορική άποψη ενδιαφέροντα. Μάλιστα, λάβαμε τα τελευταία χρόνια πολλά μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη βιωσιμότητα της αλίας. Εφαρμόζουμε τέσσερις μήνες βιολογικού πάψης παύσης, ελάχιστο όριο 500 γραμμαρίων καθαρισμένου ψαριού. Επίσης ένα δεύτερο σχέδιο χωροταξίας ε, και διαχείριση της αλίας βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης. Θα ήθελα τώρα να υποστηρίξω ότι η ευρωπαϊκές χώρες υποστηρίζουν αυτή την προσπάθεια εξασφάλιση βιωσιμότητα έλεια. Για παράδειγμα, η γαλλική, ο Γαλλικό Συνεταιρισμό, η ΕΦΔΕ, χρησιμοποίησε όλες τις μελέτες για την ε, αναβάθμιση των υγειονομικών προδιαγραφών ε, των ε, εργοστασίων μας και επίσης έγιναν δωρεέ πολλών σωσιβίων γυλαίκων ο γερμανικός συνεταιρισμός συνέβαλε και επένδυσε στην ενίσχυση του, ελέγχου και της εποπτείας. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα έχουμε διαφοροποιήσει τις δραστηριότητές μας. Επεκταθήκαμε και στην αλία Φρύσας, γιατί και ο, πολιτισμός, ο πληθυσμός της Αλίας, ο πληθυσμός συγγνώμη, της Μαυριτανίας χρησιμοποιεί και καταναλώνει ψάρι και καθημερινά. Έχει ενταχθεί το ψάρι στη διατροφή. Βέβαια για την Αλία Φρύσας πρέπει να βγούμε σε ζώνες ε, με βάθος 20 μέτρων. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, ε, πυρόγες και σκάφη βιοτεχνικά που θα είναι πιο ασφαλή και πιο στερεά για να μπορούμε να λιεύουμε σε βαθιά ύδατα. Βέβαια το, το ελευτικό απόθεμα της Φρύσας είναι κοινό με τους, με τους γείτονες της Δυτικής Αφρικής που επίσης χρησιμοποιούν στη διατροφή τους το είδος αυτό. Έχουμε λοιπόν διαπραγματεύσεις με τους παράκτους αλληλείς της Ενεγάλης και της Γκάμπιας για να δούμε πώς από κοινού θα προωθήσουμε μια κοινή διαχείριση που θα δίνει έμφαση και προτεραιότητα στην παράκτη αλληλεία μικρής κλίμακος αλλά και στην κατάκτηση των τοπικών αγορών. Αν σας εξηγώ όλα αυτά τα σχέδια που έχουμε για την ε, ανάπτυξη της βιώσιμης αλληλείας είναι γιατί εσείς οι ευρωβουλευτές θα ήθελα να καταλάβετε ε, ποια είναι τα διακυβευόμενα στην ε, εταιρική αυτή σχέση, στην αλληλευτική συμφωνία σύμπραξης, γιατί η Ευρώπη είναι και θα παραμείνει ο μεγαλύτερος εταίρος ε, σε θέματα αλληλείας, αλλά θέλουμε να είναι δίκαιος ο εταίρος αυτός. Δίνουμε μάχη για το θέμα αυτό από το 1996 και σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Γι' αυτό ήρθα και εγώ να σας μιλήσω πρόσωπο με πρόσωπο. Και θα ήθελα να σας πω το εξής. Έχουμε και τα υλικά μέσα αλλά και τους ανθρώπινους πόρους για να ε, αξιοποιήσουμε με βιώσιμο τρόπο το αλληλευτικό απόθεμα του χταποδιού και μεγάλο τμήμα των άλλων πόρων μας. Θέλουμε λοιπόν να, ε, να μας αφήσετε το χταπόδι μας. Το ίδιο μήνυμα το στείλαμε και στην κυβέρνησή μας όταν διαπραγματευόταν ε, μια σύμβαση με την Κινέζικη εταιρεία Πόλη Χοντών το 2011 μια συμφωνία που αντέβαινε στα συμφέροντα των Μαυριτανών αλλιέων. Κάναμε εκστρατεία, κινητοποιήσαμε την κοινωνία των πολιτών, τα μέσα μαζική ενημέρωσης, οργανώσαμε διαδηλώσει, συλλαλητήρια μπροστά στη, στα γραφεία της διοίκηση. Μάλιστα είχαμε αντιπαραθέσεις με τους υπαλλήλους και στη τηλεόραση, λέγοντας το ίδιο, ότι αυτό που μπορούμε εμεί να αλλιεύσουμε θα πρέπει να το αφήσουν σε εμά είναι κάτι αδιαπραγμάτευτο, είναι το μεροκάματό μας, είναι η τροφή μας, αλλά και η θέση εργασίας για τους συμπολίτε μας. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, συμφωνία με τους Κινέζους, την περασμένη εβδομάδα λάβαμε μια χαρμόσυνη είδηση. Η κυβέρνηση μας ενημέρωσε ότι οι δραστηριότητες της ε, Κινέζικης εταιρείας Χοντών... θα περιοριστεί πια στα μικρά πελαγικά είδη και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανήγγειλε σε μια συνέντευξη τύπου ότι οι όροι που θα προσέφερε στους Κινέζους και σε όλους ε, τους αλλοδαπούς στόλους θα ήταν οι ίδιοι με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα ισχύουν για τους ευρωπαϊκούς στόλους. Μάλιστα διευκρίνησε ότι το χταπόδι θα το αλλιεύουν μόνο οι Μαυριτανοί αλλιείς και μάλιστα οι Μαυριτανοί αλλιείς παράκτες αλίες μικρής κλίμακας. Αυτές οι τεχνικές διαπραγματεύσεις λοιπόν και οι τεχνικές προϋποθέσεις για τον ευρωπαϊκό στόλο βαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση κατά τη γνώμη μας μας επιτρέπει να εκμεταλλευτούμε εμείς οι ίδιοι το χταπόδι μας, βασικό στοιχείο του πρωτοκόλλου. Μάλιστα, δημιουργήθηκαν νέες ελευτικές ζώνες, κάτι που συνιστά πρόοδο. Γιατί αν αφήσουμε τις μηχανότητες να λιεύουν στην ανοιχτή θάλασσα, θα προστατεύσουμε καλύτερα το βυθό. Θα μειώσουμε τα, τα παραλιεύματα και θα μειώσουμε και τα, και τα ατυχήματα με τις βιοτεχνικές πυρόγες. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχετε υπόψη σας ότι το μισό ελευτικό ε, ε, απόθεμα της ε, τσιπούρας μας είναι παραλίευμα ουσιαστικά των μηχανότρατων που αλλιεύουν φρύσα. Δεν είναι δυνατόν έτσι να εξασφαλίσουμε βιώσιμη αλληλεία. Τι θέλετε να κάνουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα την χρηματική αντιπαροχή, τη χρηματική αντιστάθμιση. Για το πιο σημαντικό δεν είναι να έχουμε ένα δέκα εκατομμύρια, εκατό εκατομμύρια ευρώ. Είναι το θέμα να αξιοποιηθούν αυτά τα κονδύλια και μάλιστα με διαφωνή τρόπο για να προωθηθεί η ανάπτυξη στη Μαυριτανία. Η διαφάνεια στον τομέα της αλίας, είτε για τη χρήση ε, των κονδυλίων ε, για την αλία, είτε για τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας είναι για μας απαραίτητο στοιχείο. Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίξαμε την συμπερίληψη της αλίας στην πρωτοβουλία ε, διαφάνειας των εξορυκτικών βιομηχανιών, ITEIE. E. Είναι η πρώτη φορά που ε, μια χώρα, η Μαυριτανία προκειμένου, θέλει να εντάξει και την αλία της αυτή την πρωτοβουλία διαφάνειας. Γίνονται πολλές προσπάθειες από το αρμόδιο υπουργείο. Σε ό,τι αφορά τη χρησιμοποίηση ε, της χρηματικής αντιπαροχής των συμφωνιών, εμείς οι παράκτη αλείς ε, εκφράζουμε τη λύπη μας γιατί δεν είδαμε ούτε ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι αφορά τις επενδύσεις στις υποδομές μας. Ούτε σε ό,τι αφορά τη μεταφορά τεχνογνωσίας στα λιμάνια, στα εργοστάσια μεταποίησης, ε, ε στη, στις αποθήκες, στα προγράμματα κατάρτισης και ούτω καθεξής τέτοιες επενδύσεις θα είναι πολύ σημαντικές και χρειάζονται αν θέλουμε να έχουμε μια πραγματικά εταιρική σχέση που θα είναι επωφελής για όλες τις πλευρές. Αυτό ελπίζουμε να γίνει στα πλαίσια του νέου πρωτοκόλου. Και επίσης ε, προσβλέπουμε στην υποστήριξή σας γι' αυτό. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Αχμέτ. Α, ε, διακόπτη ο μιλητής. Δυστυχώς Ξεχάσαμε προηγουμένως να φωτοτυπήσουμε το κείμενο, αλλά στο μεταξύ έχει ολοκληρωθεί η, φωτοτυπή, η φωτοτυπήση. Μπορείτε να λάβετε τα αντίγραφα στην είσοδο της αίθουσα. Ωραία. Τώρα περνάμε στον τελευταίο μας ομιλητή, κύριο Χαβιέρ Γκαράτ, τον πρόεδρο της ε, ε, Ευρωαλίας, Ευρωπέσκα. Έχετε το λόγο κύριε Γκαράτ. Σας ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ως πρόεδρος της Ευρωπές ε, θα μιλήσω για την υπόλοιπα είδη, γιατί ο συνάδελφος, ο, ο πρώτος ομιλητής μίλησε για τα πελαγικά είδη. Το πρώτο σχόλιο είναι ότι η διαπραγμάτευση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, καθ' όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης αυτής θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως πολύ κακή διαπραγμάτευση. Αυτή είναι η γνώμη των αλλιέων. Και μάλιστα αυτό διαπιστώθηκε η κακή της ποιότητα γιατί το αποτέλεσμα δεν ήταν ε, ε θετικό για τα περισσότερα αλλιευτικά είδη. Και μάλιστα ε, λίγο πριν ε, την παρουσίαση της συμφωνίας αυτής, ε, Σίσο Μιαλής και της Μαυριτανίας και η Αλοδαπή είπαν ότι είναι καλύτερα να μην υπογραφεί συμφωνία, να μην έχουμε καν συμφωνία από το να έχουμε μια κακή συμφωνία. Έγινε, διαπραγμα... Έγινε διαβούλευση με την αρμόδια επίτροπο, ε, μας αγνώρισε και είπε ότι όσο αυτή είναι επίτροπος θα υπογραφεί η συμφωνία. Οπότε η πρώτη απορία είναι, είναι καλή ή κακή η συμφωνία. Η απάντηση είναι φως φανάρι κατά τη γνώμη μου. Ιδιαίτερα μετά από ένα εξάμεινο εφαρμογής της συμφωνίας, παρόλο που είναι προσωρινή, διαπιστώνουμε ότι είναι κακή. Έχουμε σαφή υποχρησιμοποίηση σχεδόν όλων των κατηγοριών αλληλείας και αργότερα θα σας δώσω περισσότερες πληροφορίες. Με εξαίρεση τα των αλληλευτικά και τις μηχανότρατες ψυγεία που δεν έχουν αλλάξει τεχνική όρη, ε, και μερικά παραγατιάρικα βυθού και μερικά βεθοπελαγικά, για τα υπόλοιπα είδη, για τα κεφαλόποδα που αποκλείστηκαν, αλλά και για τα πελαγικά είδη, δεν χρησιμοποιείται παρκώς συμφωνία. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ε, απώλεια εκα... χιλιάδων θέσεων απασχόλησης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Μαυριτανία. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, για τα, κεφαλοπο... για τα κεφαλόποδα και για τα ε, θαλασσινά, 35 ε, 35 πλοία έμειναν εγκυροβολημένα, 400, 400 μέλη του πληρώματος αποκλείστηκαν από την Αλία. Στα Κανάρια απολύθηκαν 1.200 εργαζόμενοι και θα φτάσουν τους 3.000. Έκλεισαν 20 επιχειρήσεις ανακοινώθηκαν 15 ε, αναδιαρθρώσεις και θα χαθούν 15 εκατομμύρια τζίρος μόνο από τα Κανάρια νησιά. Στη Μαυριτανία είχαμε εκατοντάδες ναυτικούς αλλά και προσωπικού εδάφους βρίσκονται σε ανεργία αυτή τη στιγμή και δεν, υπάρχουν, δεν έχουν καμία δυνατότητα να βρουν θέση απασχόλησης. Είναι κακή συμφωνία αυτή λοιπόν, γιατί οι τεχνικές προϋποθέσεις και οι οικονομικές προϋποθέσεις για, τις περισσότερες, για τα περισσότερα ιδεαλίες δεν είναι βιώσιμες. Παρόλο που ακόμη και τότε κατά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων οι επιχειρήσεις ήταν στο όριό τους ό,τι αφορά την, την κερδοφορία τους, Τώρα έχουμε ακόμη χειρότερα αποτελέσματα. Αν ξεκινήσουμε με την αλληλεία θαλασσινών, το κόστος άδειας έχει αυξηθεί, έχει πενταπλασιαστεί μέσα σε λίγα χρόνια. Τώρα, το τελευταίο, τελευταίο μόνο χρόνο έχει διπλασιαστεί. Ένα μέσο σκαφο ένα μεσό σκαφο θα πληρώνει 56.000 ευρώ το χρόνο, από 56.000 ευρώ το χρόνο μάλλον θα χρειαστεί να πληρώνει 127.000 ευρώ το χρόνο, δηλαδή 75.000 ευρώ το χρόνο ε, επιπλέον για τι αλληλευτικέ άδειε. Στι αλληλευτικέ ζώνε και εκεί υπάρχουν κάποιε αλλαγέ. Στο Νότο χάσαμε Πέρασαμε στην απαγόρευση από 6-8 μίλια με εξαίρεση το 50% του στόλου με ανώτατο όριο 10 πλοία. Αλλά πρώτα απ' όλα χάσαμε μια πολύ σημαντική ζώνη στο βορρά. Με βάση τα στοιχεία που μας έδωσε το Ισπανικό και ο Αναγραφικό Ινστιτούτο, θα έχουμε μια απώλεια 21,6% των αλλιευμάτων καραβίδας. 21% στο βορρά, στο βορρά και 14,6% στο νότο. Οπότε 120 120.000 ευρώ το χρόνο λιγότερα έσοδα. Επίσης, ε, είχαμε συμφωνία για 50.000 ε, τόνους, για ένα πληθυσμό όμω που θέλει βιώσιμη αλεία και αηφόρα αλεία και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος ε, υπερεκμετάλλευσης. Μάλιστα δεν υπάρχουν καν ε, επιστημονικά πορίσματα που να ζητάν τάκ. Το να επιβάλλεται τάκ, κατά τη γνώμη μας, είναι απαράδεκτο. Σε ό,τι αφορά τα παραλιεύματα, τα bycatch. 15% ε, για στα κεφαλόποδα έχει απαλληθεί. Οπότε μειώθηκαν από 20% σε 10% τα παραλιεύματα, οπότε θα έχουμε αντίκτυπο 36.000 ε, ευρώ για κάθε ε, πλοίο και από 26% σε 5% για τα καβούρια. Πέρα λοιπόν της, του οικονομικού αντικτύπου θα έχουμε και ε, ενίσχυση των απορρίψεων γιατί θα χρειαστούν να απορρίπτουν τα παρελίευματα. Σε ό,τι αφορά την κατηγορία 2, μηχανότρατες, όχι ψυγεία και επίσης αλία μαύρου μερλούκιου. Εκεί έχει αυξηθεί αισθητά ε, από 250 σε 350 ε, η κιορτή. Επίσης δόθηκε τάκ 400 ε, Χωρί χωρίς ε, επιστημονική αιτιολόγηση. Μόνο δύο είναι τα σκάφη αυτή τη στιγμή και αυτά τα δύο σκάφη κατά πάσα πιθανότητα θα το αλλιεύαν σε λιγότερο από ένα χρόνο και επίσης διευρύνεται ε, η απαγόρευση από 6 στα 8 μίλια, κάτι που θα έχει επίσης αντίκτυπο. Σε ό,τι αφορά τα σκάφη που, που αλλιεύαν ε, κεφαλόποδα, γιατί, όπως είπα, για τα τοναληφτικά δεν έχουν αλλάξει τεχνικές προϋποθέσεις. Θα συνεχιστεί η χρησιμοποίηση της συμφωνίας. Τώρα, κατηγορία 9, κεφαλόποδα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ένα ψήφισμα του Μαΐου του 2011 είπε ότι υπήρχε υπερεκμετάλλευση των κεφαλόποδων. Μπορούμε να δηλώσουμε σήμερα ότι οι επιστημονικές πληροφορίες που υπάρχουν για το αλίευμα, για το ληφτικό απόθεμα των κεφαλοπόδων οδηγήσει στο αντίθετο συμπέρασμα. Είναι εσφαλμένη αυτή η δήλωση για υπερεκμετάλλευση και μάλιστα το Ισπανικό Κοινογραφικό Ινστιτούτο έχει συγκεντρώσει στοιχεία 300.000 ε, στοιχεία και 8.000 δείγματα από χταπόδι δείχνουν ότι η κατάσταση του αποθέματος χταποδίου τελευταία 25 χρόνια είναι άριστη και μάλιστα και η ΕΤΟΕΑ ε, κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα αλλά δυστυχώς δεν χρησιμοποιήθηκε η δική της μελέτη παρά οι μελέτες των προηγούμενων ετών, 2008-2009, για ένα είδος αλλιευτικό που μέσα σε ένα χρόνο πεθαίνει, είχε μόνο ένα έτος κύκλο ζωής. Είναι σαφές λοιπόν ότι ήταν ανακριβείς και ακατάλληλες αυτές οι επιστημονικές πληροφορίες. Μάλιστα τον Ιούλιο του 2012 ο σκάφο, το αλληλευτικό στόλος είχε αποδώσει πάνω από το 300% με βάση τα στοιχεία του Μαυριτανικού και Ονογραφικού Ινστιτούτου. Έχει μειωθεί λοιπόν ο, κατά 55 πλοία ο ελευτικός στόλο, από 55 το 2011, 2001 συγγνώμη λέει ο σε 31 σκάφη το 2012. Οπότε τηρήθηκε το σχέδιο διαχείρισης του χταποδιού και των κεφαλοπόδων στη Μαυριτανία. Ελάχιστη ήταν από τις ελάχιστες περιπτώσεις που είχαμε εφαρμογή πραγματική του σχεδίου διαχείρισης από τον ελευτικό στόλο. Δεύτερη ε, απορία. Είναι προσοδοφόρα αυτή η συμφωνία. Ε, δηλαδή πιάνουν, κόπο τα χρή... τόπο τα χρήματα, αξίζει τον κόπο. Πιστεύω ότι είναι πολύ δαπανηρή. 70 εκατομμύρια ευρώ για λιγότερες αλληλευτικές δυνατότητες, Τα κεφαλόποδα αποκλείονται. Δεν μειώθηκε μάλιστα η χρηματοοικονομική αντιστάθμιση, η αντιπαροχή, παρόλο που στα προηγούμενα πρωτόκολλα και η συμπερίληψη των κεφαλοπαιόδων και ε, με την συμπερίληψη των πελαγικών αυξήθηκε η χρηματική αντιπαροχή. Στην περίπτωση των θαλασσινών έχουμε μείωση κατά 21%, ακόμη και αν έχουμε προσοδοφόρα αλία, μειώνεται κατά 21% η αλία. Ε, το μερλούκι έχουμε το νότο όριο των 300.000 που έχει μπει νέα τάκ. Επίσης έχει αυξηθεί από 200 σε 300% το άλλο είδος. Βέβαια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται επαρκώ τα κονδύλια, το, τα χρήματα των φορολογουμένων να πιάνουν τόπο. Αλλά αυτό θα πρέπει να ισχύσει και στην Ελευτική Συμφωνία. Είναι πιο βιώσιμη η τελευταία συμφωνία από τι προηγούμενε. Όχι, ούτε από οικονομική, ούτε από κοινωνική άποψη και δώσαμε τι αποδείξει. Τώρα, από περιβαλλοντική άποψη. Οι νέε ζώνε προστατεύουν τα οικοσυστήματα. Εμεί θεωρούμε ότι καλύτερη ε, επιστημονική γνώση και οι πρόσφατες γνώσεις επιστημονικές δεν χρησιμοποιήθηκαν. Για τα κεφαλόποδα, για παράδειγμα, τα τάκ για το μαύρο μαλλούκιο και τα θαλασσινά. Και επίση ο περιορισμό τη αλληλευτική ζώνη δεν χρησιμοποιήθηκε με βάση κανένα αντικειμενικό επιστημονικό κριτήριο. Για τα θαλασσινά, η ζώνη που χρησιμοποιήθηκε, αυτό που λένε οι ε, ε, οι μελέτες λένε ότι δεν γίνεται ελεία σε ευαίσθητα οικοσυστήματα, σε ευαίσθητους βυθούς, αλλά σε αμμόδι βυθό που δεν είναι καθόλου ευαίσθητος από περιβαλλοντική άποψη. Τώρα, οι ζώνες που αλλιεύουν τα δικά μας σκάφη δεν έρχονται σε σύγκρουση ε, συμφερόντων με τα μαυριτανικά σκάφη. Ε, ο στόλος μας δυστυχώς θα χάσει πολύτιμες ε, επιστημονικές πληροφορίες γιατί στους στόλους θαλασσινών είχαμε μονίμως έναν εμπειρογνώμονα που συνέλεγε στοιχεία. Και μην ξεχνάμε ότι αν φύγουμε εμείς από, από τη Μαυριτανία θα μπουν άλλες χώρες και θα λιεύουν που δεν έχουν τόσο υψηλές προδιαγραφές όπως οι Κινέζοι για παράδειγμα. Τώρα για την εκφόρτωση στη Μαυριτανία. Εμείς προτιμούσαμε το προηγούμενο σύστημα. Να είναι προαιρετικό ε, για την εκφόρτωση για όσους είχαν τέτοια δυνατότητα. Γιατί, μεταξύ άλλων, επειδή έχουμε ε, ε, τα Κανάρια νησιά, που είναι εξόχως ε, απόκεντρη περιφέρεια, με τεράστιες επιδράσεις ό,τι αφορά την απώλεια θέση απασχόλησης. Όπως σας είπα και πριν, ήδη απολύθηκαν 1.200 άνθρωποι και θα φτάσουν οι απολύσεις στις 3.000. Επίσης θα μπουν σε εφαρμογή 15 συστήματα αναδιάρθρωσης. Και μην ξεχνάμε και το νομικό σύστημα για τις εξόχως τις περιοχές. Θέλουμε συνέπεια μεταξύ των αποφάσεων και των εφαρμογών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των όρων συμφωνιών με τρίτες χώρες, ώστε να μην φέρουμε σε δυσμενή θέση τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, εμπροκειμένου τα Κανάρια νησιά. Θέλουμε να είναι επαφελής συμφωνίες και για τις δύο πλευρές, εμπροκειμένου για τη Μαουριτανία, αλλά και για, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ για τις Κανάριες νήσους. Τώρα, ο νέος τρόπος υπολογισμού είναι καλύτερος? Όχι, γιατί ε, δίνεται λαβή για διαφθορά και για αδικαιολόγητες οικονομικές κυρώσεις που αφορούν το ζήγισμα των αλλιευμάτων στον τόπο ελέγχου είχαμε τέτοια παραδείγματα στο παρελθόν, θα τα έχουμε και στο μέλλον με τον νέο υπολογισμό. Το πρωτόκολλο είναι μη βιώσιμο και από τεχνική και από οικονομική άποψη για τα περισσότερα αλλιευτικά είδη. Θα είναι πολύ δαπανηρή συμφωνία. Θα πληρώσουμε 70 εκατομμύρια στη Μαυριτανία για δυνατότητε αλλίε που υπό τι τρέχουσε συνθήκε δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Δημιουργούνται τεράστια οικονομικά και κοινωνικά μειονεκτήματα. Θεωρούμε ότι θα πρέπει επιγόντω να συνεδριάσει η Κοινή Επιστημονική Επιτροπή για να δώσει την τελευταία της εκτίμηση για το χταπόδι και τα άλλα είδη, δηλαδή να συνέλθει η Μεικτή Επιτροπή και να συζητηθούν όλα τα προβλήματα και για το πελαγικό στόλο και για τα υπόλοιπα είδη. Αλλιώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το άρθρο 5 του πρωτοκόλου και να καταγγείλει για εμφανή υποχρησιμοποίηση των ελληνικών συμφωνιών ε, δυνατοτήτων και να ζητήσει νέα διαπραγμάτευση του πρωτοκόλου. ΔΕΜΗ, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει το πρωτόκολλο, να μην το κυρώσει, ζητώντα από τα ενδιαφερόμενα μέρη κατεπηγόντω να διαπραγματευτούν νέο πρωτόκολλο. Γιατί αυτό που θέλουμε είναι να λιεύουμε υπό πρόσφορε συνθήκε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ του τέσσερι εμπειρογνώμονέ μα για τι παρουσιάσει του και τώρα θα έχουμε μία ανταλλαγή απόψεων, ένα γύρο έρωτα απαντήσεων. Η κυρία Λεβίν ζήτησε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που έφτασα καθυστερημένη. Καθυστέρησε η πτήση μου, δυστυχώς. Αυτός είναι ο λόγος. Και ζητώ συγγνώμη και από τους εμπειρογνώμονε που δεν τους άκουσα. Δεν είχα τέτοια πρόθεση. Έχω κάποιες ε, ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα τον κύριο Γκαρά που μόλις τώρα αναφέρθηκε στο Ισπανικό και Οκεανογραφικό Ινστιτούτο και τα πρόσφατα πορίσματά του και αναφέρθηκε επανειλημμένα στην έκθεση. Από ό,τι γνωρίζω, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι η ίδια έκθεση που παρουσιάστηκε στην, στην συνεδρίαση στις Βρυξέλλες. Τίτλος «Ταχεία αξιολόγηση των αποθεμάτων του χταποδιού και του ε, μπακαλιάρου της Ενεγάλης. Ο συγγραφέας της εκθέσεως ήταν προσεκτικός και είπε ότι δεν ήταν πλήρης η αξιολόγηση και εμπεριείχε κάποιες ε, ενδείξεις για ανάκαμψη του αποθέματος αν ακολουθούνται κάποιες συστάσεις και αν ήταν ευνοϊκές οι περιβαλλοντικές συνθήκες. Θέλω να ακούσω περισσότερα για τη μελέτη. Ανορίζει ο κύριο Γκαράντ ότι η τρίτη χώρα μπορεί να εκτιμήσει το πλεόνασμά της. Αν η Μαυριτανία έχει στρατηγική για την ανάπτυξη της δικής της αλίας, όπως ακούσαμε να μας λέει ο κ. Σινταμέντ, ο πρόεδρος της Ενώσεως Αλιέων ε, Μικρής Κλίμακος που εκπροσωπεί 36.000 αλλήλει. Ε, θα πρέπει να αφήσουμε τη Μαυριτανία, την εξάρτητη χώρα, να πάρει την κατάλληλη απόφαση. Τον πρώτο εμπειρογνώμονα δεν τον άκουσα. Ο κ. Μπενουά. Ε, αναφέρθηκε στην αξιολόγηση. Ποιος είναι ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος του ευρωπαϊκού στόλου και δικαιολογείται η απομάκρυνσή τους από τις ακτές όσον αφορά τη συνέπεια που έχει αυτό για τα παρελιεύματα και το πώς επηρεάζει το βυθός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να απαντήσει πόσα πλοία χρησιμοποιούν εφαρμόζει το πρωτόκολλο σε αυτή τη φάση. Υποχρησιμοποιείται πόσα σκάφη εφαρμόζουν το πρωτόκολλο σε αυτή τη φάση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρώτα θα ακούσουμε τις ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών και μετά θα δώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονες, γιατί ίσως ε, ε, υπάρξει επικάλυψη και μεταξύ των ερωτήσεων. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Φράγκα. Ευχαριστώ τους καλεσμένους για τις παρουσιάσεις τους. Κάτι που προέκυψε με σαφήνεια είναι ότι η διαπραγμάτευση δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Ούτω ή και την προηγούμενη συμφωνία δεν είχαμε επικρίνει για του ε, τεχνικού όρου και προποθέσει κάποιων αλληλευτικών ειδών και εκεί είχαμε μεγάλη εκμετάλλευση ό,τι αφορά τα κεφαλόποδα, τα θαλασσινά και τις πελαγικές μηχανότρατες. Ήταν ήδη λοιπόν και η προηγούμενη αλληλευτική συμφωνία κακή και υποτίθεται ότι αυτές οι κατηγορίες δικαιολογούσαν την υψηλή αντιπαροχή και αυτά τα ίδια όμως έμειναν έξω της, εκτός της νέας συμφωνίας. Τα κεφαλόποδα, ε, αποκλείστηκαν. Σε ό,τι αφορά τις μηχανότρατες ε, για τα πελαγικά είδη και τα σκάφη ε, που ελίβα θαλασσινά, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις τεχνικές προϋποθέσεις. Οπότε, θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει γιατί πληρώνουμε τόσο μεγάλη αντιπαροχή για μια ληφτική συμφωνία που δεν χρησιμοποιείται. Και για να απαντήσω στην κυρία Λοβέν, θα ήθελα να πω ότι έχουμε δύο σκάφη αλίας μαύρο μερλούκιο, τέσσερα παραγαδιάρικων βυθού και δεν ξέρω αν έχουμε ε, μία πελαϊκή μηχανότρατα που σκέφτεται να πάει, γιατί είναι σχεδόν απεγνωσμένη η κατάσταση. Βλέπετε λοιπόν ότι η κερδοφορία είναι μηδενική Ελάχιστα είναι τα πλοία που αλλιεύουν. Ναι, για τα τοναλευτικά ισχύει, αλλά ο τόνο αποδίμησε προ άλλε ζώνε. οπότε τα τοναλευτικά ουσιαστικά, από τα έχουν μείνει δύο παραγαδιάρικα που αλλιεύουν τόνο. Οπότε ελάχιστη χρησιμοποίηση τη αλλιευτική συμφωνία και από ό,τι ξέρω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη έχει καταβάλει τα πρώτα 70 εκατομμύρια ευρώ στη Μαυριτανία. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την κατάσταση των αλλιευτικών αποθεμάτων. Και εκεί έχω πολλέ ερωτήσει. Αναφέρθηκε ρητά από τον κύριο Καγιάρ, τον πρώτο καλεσμένο, ότι στην τελευταία μελέτη έχουμε στοιχεία του 2009, είναι η μελέτη του 2010, ενώ ε, τα στοιχεία του Ισπανικού Οκεανογραφικού Ινστιτούτου μιλούν για πιο πρόσφατα χρόνια, 2011. Άλλωστε πρόκειται για μια μελέτη που μετά από αυτά που είπε ο κύριος Καγιάρ ε, δείχνει με μεγαλύτερη σαφήνεια την κατάσταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει την πιο πρόσφατη μελέτη. Αντίθετα, θα ήθελα να ρωτήσω τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρείτε ακόμη ότι η κατάσταση των κεφαλοπόδων είναι κακή, ενώ οι τελευταίες επιστημονικές μελέτες, οι πιο πρόσφατες επιστημονικές μελέτες των ωκεανογραφικών Ινστιτούτων, όχι μόνο του Ισπανικού, δείχνουν ότι η κατάσταση του ελευτικού αποθέματο των κεφαλόποδων είναι μια χαρά. Ε, λένε ότι αν δεν έχουν πλεονάσματα οι Μαυριτανοί δεν μπορούμε εμείς να αλλιεύσουμε. Μα υπάρχουν και πλεονάσματα. Οπότε περισσεύουν και για τον Ευρωπαϊκό Αλλιευτικό Στόλο. Σε ό,τι αφορά την παράκτη αλία της Μαυριτανίας, ερωτώ, γίνεται σε ζώνες όπου αναπαράγεται το χταπόδι, γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν προβληματικό, αν υπάρχουν και γόνοι χταποδιού. Σε ό,τι αφορά τώρα τα σκάφη αλίας θαλασσινών. Γιατί προσδιορίστηκαν κάποιες αλλιευτικές ζώνες ενώ το απόθεμα είναι βιώσιμο. Μάλιστα γίνεται σε αμμώδεις βυθούς, δηλαδή δεν βλάπτει το οικοσύστημα, γιατί επαναλαμβάνω η βυθή είναι το ενώ ταυτόχρονα η ζημία που προκαλεί στον κλάδο είναι τεράστια που ούτως ή άλλως ήταν οριακή η κατάσταση του κλάδου των θαλασσινών. Και μάλιστα μόλις σε πλέον υποχρέσεις που δημιουργεί η συμφωνία θα έχουμε 33% μείωση των εσόδων, για να, ζημιών μάλλον των σκαφών αλίας θαλασσινών. Πώς θα τολμήσουν λοιπόν ε, να πάνε οι Ευρωπαίοι αλίες να αλλιεύσουν θαλασσινά εκεί με τέτοιες ζημιές. Θα ήθελα να υποβάλω μια ερώτηση και στον εκπρόσωπο της Μαυριτανίας. Η παράκτια αλία μικρής κλίμακος της Μαυριτανίας απαρτίζεται από Σενεγαλέζους, αν δεν κάνω λάθος αλίες. Η πλειοψηφία είναι Σενεγαλέζοι, δεν είναι καν Μαυριτανοί. Το επιβεβαιώνετε, γιατί μας μίλησε για 36.000 ψαράδες ε, αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι είναι Σενεγαλέζοι και όχι Μαυριτανοί. Ενώ ο αντίκτυπος που θα έχουν τα μέτρα αυτά στο λιμάνι του Αντιμπού θα επηρεάσουν χιλιάδες μαυριτανούς ψαράδες ή ε, ανθρώπους που απασχολούνται στην Αλία. Θα έχει τεράστια επίδραση λοιπόν στο, στην Αλία της Μαυριτανίας. Και αυτό το κοινωνικό θέμα θα είναι αισθητό και στην Ευρώπη δεν ε, περιοριζόμαστε μόνο στο λιμάνι του Μαριμπού. Εκεί πραγματικά οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες είναι πολύ σημαντικές και αρνητικές εννοώ. Πιστεύω ότι και μία ακόμη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύτηκε τεχνικές ε, προϋποθέσεις που δεν έχουν καμία σχέση με τις αλληλευτικές δυνατότητες. Και ένα άλλο παράδειγμα, το θέμα του Μαύρου Μερλούκιου. Εκεί η διαπραγμάτευση έγινε για 11 σκάφη και για τα 4.000 τόνους ε, ανώτατη ποσόστοση, που φτάνει το πολύ για δύο σκάφη. Γιατί δύο είναι τελικά τα σκάφη που αλλιεύουν εκεί όπως ε, διαπιστώνουμε. Γιατί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύτηκε ε, πράγματα που είναι τελείως ανέφικτα να εφαρμοστούν. Και τέλος, όταν ο τομέας και οι εθνικές διοικήσεις που εκπροσωπούν τον τομέα λένε όλες είναι απαράδεκτη συμφωνία, θα πρέπει για επιτέλους να έρθει η Επιτροπή να μας εξηγήσει γιατί ε, υπέγραψε μια συμφωνία που υπό αυτές τις συνθήκες δεν τη θέλει κανένας. Ευχαριστώ. Να δώσω τώρα το λόγο στον επόμενο μιλητή. Απευθύνονται ερωτήσεις και προς τους καλεσμένους και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά επαναλαμβάνω σε αυτή τη φάση της συζήτησης να υποβληθούν ερωτήσεις μόνο προς τους εμπειρογνώμονές μας. Στη δεύτερη ενότητα. Όταν θα σα παρουσιάσω εγώ την έκθεσή μου, κυρία Φράγκα, θα υποβάλουμε ερωτήσει και προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή σε αυτή την ενότητα, παρακαλώ, περιοριστείτε μόνο σε ερωτήσει προ του εμπειρογνώμονέ μα. Ο κύριο Αρσένη. Uh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι είναι λογική αυτή η συμφωνία για ένα λόγο, αν μη τι άλλο ακολουθεί αυτά που ζητήσαμε στο ψηφισμά μας. Πώς θα πρέπει να συντάσσονται αυτές οι συμφωνίες για τη χείριση του, των ελευτικών αποθεμάτων. Για πρώτη φορά εφαρμόζονται οι αλλαγές που ζητήσαμε στις νέες αλληλευτικές συμφωνίες. Για πρώτη φορά εφαρμόζεται αρχή ότι πρέπει να λιεύεται το πλεόνασμα ανέφερε κύριε Φράγκα από θέματα που δεν μπορούμε να τα εκμεταλλευόμαστε πλέον. Επειδή είχαν υπεραλλιευθεί. Συμβαίνει αυτό και μόνο με αλίευση του πλεονάσματος μπορούμε να αποκαταστήσουμε τα αποθέματα και να δώσουμε ευκαιρίες στους αλείς των χωρών αυτών ε, να αλλιεύουν ε, όλων των χωρών του πλανήτη. Ακολουθούμε σωστό δρόμο. Είναι λογικό το ότι στην πρώτη φάση πρέπει να πληρώσουμε το τίμημα για τις ζημιές που σημειώθηκαν. Τα αλλιεύματα θα είναι μικρότερα. Αυτό γιατί επιλέξαμε τη βιωσιμότητα. Να μην έχουμε περισσότερα, για να έχουμε περισσότερα πλεονάσματα και περισσότερη αλήψη στο μέλλον. Ευχαριστώ, κυρία Μπιλμπάου. Ευχαριστώ. Με κάλυψαν οι συνάδελφοι σε πολλές ερωτήσεις. Θα ήθελα όμως, ε, σε σχέση με τις μελέτες που λένε ότι το απόθεμα χταποδιού βρίσκεται σε, καλές, ε, σε καλή κατάσταση, θα ήθελα να ρωτήσω τους εμπειρογνώμονές μας τι γνώμη έχουν. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν χρησιμοποιήσει αυτό το στοιχείο. Μπορούν να μου πούνε οι εμπειρογνώμονες αν ε, έδωσε σε εκείνους τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξήγηση για το ότι αγνόησε αυτή την πληροφορία των μελετών ότι το απόθεμα χταπόδιου είναι σε καλή κατάσταση. Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν μέχρι και πλεονάσματα και μάλιστα η Μαυριτανία μπορεί να αποφασίσει να χρησιμοποιήσει αυτούς τους πόρους για τον δικό της αλληλευτικό κλάδο. Θα ήθελα λοιπόν εκπρόσωπος ε, των ε, Μαυριτανών ψαράδων να μου πει έγινε μια αξιολόγηση της ζημίας που μπορεί να έχει όχι μόνο στον τοπικό πληθυσμό από την έλλειψη αλληλευτικών αδειών για τα ευρωπαϊκά σκάφη, αλλά τι γίνεται με την κατάρτιση των τοπικών πληθυσμών, των ντόπιων ε, για εργασία σε πλοία και ούτω καθεξής. Όλοι ξέρουμε ότι τα αλληλευτικά εξάντλησαν πέρυσι τις αλληλευτικές άδειες, χρησιμοποίησαν και φέτος ε, επίσης θα έχουν. Πρέπει να καταβάλουμε όμως προσπάθεια για να καλύψουμε τις ανάγκες του κλάδου. Γιατί όπως ακούσαμε και ο ελευτικός κλάδος είναι κατά της ελευτικής συμφωνίας. Γιατί φαίνεται ότι δεν επικερδίζει τελικά αυτή η συμφωνία για κανέναν. Δεν έχει νόημα να συνεχίσουν την αλληλεία στα ύδατα της Μαυριτανίας. Έχω και ερωτήσει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα τις υποβάλω στη δεύτερη ενότητα. Ευχαριστώ. Κύριος Ρωμέβα. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση θα ήθελα μόνο να υποβάλω μετά από αυτές που έθεσε και η κυρία Λεβίν. Μία ερώτηση για τον κύριο Σίνταρ Αχμέτ. Μήπως κάνετε ένα μικρό υπολογισμό για το πόσες θέσεις εργασίας θα προκύψουν αν η διαχείριση του χταποδιού γίνεται απευθείας από τους μαυριτανούς ψαράδες. Μόνο αυτό θα ήθελα να ρωτήσω. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Άγνιο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα. Χιόνιζε στη Βρετανία και φαίνεται ότι πλήττει το μεταφορικό σύστημα στη Βρετανία. Um, Δεν άκουσα αυτά που είχε να πει ο κύριος από τη Μαυριτανία. Βλέποντας αυτές τις σημειώσεις, εκφράζοντας τη βρετανική άποψη, κάτι που πάντα θα κάνω εδώ, Λέγω ότι θεωρώ ότι είναι και καλυμμένη ε, εξωτερική ενίσχυση. 70 εκατομμύρια ευρώ πληρώνει ο Βρετανός ε, φορολογούμενος που δίδονται στη Μαυριτανία και επιτρέπεται περισσότεροι σε Νεγαλέζοι αλείς να ψαρεύουν εκεί. Μάλλον, άμα το δει κανεί κοινικά έτσι είναι. Με διαβεβαιώνεται ότι το βρετανικό στοιχείο, τα 70 εκατομμύρια, πραγματικά θα βοηθήσει τον λαό της Μαυριτανίας. Ευχαριστώ. Gracias, señor Ευχαριστώ, ο κύριος Σάντζες Πρεσέδο. Ευχαριστώ. Μόνο ερωτήσεις τώρα, έτσι, επί της ουσίας αργότερα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας δείξω εδώ ένα περιοδικό της 31ης Δεκεμβρίου από τη δική περιφέρεια που κάνει μια σύνοψη της αλίας στη Γαλλικία. Ε, ο τίτλος είναι «Η Γαλλική λέει αντίο στη Μαυριτανία». Ερωτώ λοιπόν τον κύριο Καγιάρ. Έγινε ένας υπολογισμός του κοινωνικού αντικτύπου της συμφωνίας αυτής. Ε, τα στοιχεία που έλαβε υπόψη συμφωνία είναι για το 2008 και το 2009. Γιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν μεταγενέστερα πιο πρόσφατα στοιχεία. Θα έπρεπε να επαναξιολογηθεί δεδομένη της νέας κατάστασης του αποθέματος χταποδιού. Σε ό,τι αφορά την ενδιαφέρουσα παρουσίαση που είχαμε από τον Μαυριτανό Ψαρά και πρόεδρο του Μαυριτανικού Συνεταιρισμού. Η ΕΤΟΕΑ μίλησε και για άλλους ε, στόλους που αλλιεύουν κεφαλόποδα. Ισχύει αυτό. Υπάρχουν και ελευτικοί στόλοι άλλων κρατών που αλλιεύουν κεφαλόποδα στα χωρικά ύδατα της Μαυριτανίας γιατί η Επιστημονική και Οικονομική Επιτροπή ζήτησε αποτίμηση του διαλόγου για του αντικτύπου για την υποχρέωση εκφόρτωσης, τον αντίκτυπο που θα έχει αυτή η υποχρέωση εκφόρτωσης στον τοπικό πληθυσμό. Έχετε σχετικές πληροφορίες. Κύριε Χαβιέρ Γκαράτ, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Πιστεύετε ότι μπορούμε να κάνουμε κάποιες διορθώσεις ή κάποια αναθεώρηση του πρωτοκόλλου μετά την υπογραφή ώστε να γίνει πιο υποφερτό ή θεωρείτε ότι χρειαζόμαστε αναδιαπραγμάτευση μια εκ νέου δηλαδή διαπραγμάτευση του πρωτοκόλλου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τόμας, η κυρία Τόμας, συγγνώμη. Oui, merci, Ευχαριστώ. Τα επιχειρήματα και των μεν και των δε είναι εύλογα και θεμητά. Δηλαδή έχουμε τις εύλογες απαιτήσει για ανάπτυξη των μαυριτανών αλλιέων, αλλά έχουμε ταυτόχρονα και το συναγερμό που κρούν οι Ευρωπαίοι αλληλείς ό,τι αφορά τις απολύσεις, την κατάργηση θέσεων απασχόλησης και την ανεργία των αλλιών που έμειναν στην ξηρά τους τελευταίους μήνες. Όλα αυτά εξαιτίας ε, της συμφωνίας που υπάρχει σε ό,τι αφορά την κατάσταση του αποθέματος κεφαλόποδων. Και βλέπουμε πόσο σημαντική είναι η σωστή αξιολόγηση και αναφυσβήτητα αντικειμενικά στοιχεία για την κατάσταση του αποθέματος αυτού. Γιατί αυτή η συμφωνία που υπάρχει για το χαρακτηρισμό του αποθέματος ε, συμβάλλει στην ε, ε, διαφωνία μας για το χαρακτηρισμό της ίδιας ελευτικής συμφωνίας. Θέλουμε μια συμφωνία που είναι, να είναι καλή για όλους. Επίσης, όπως είπε και η Σαμπέλα Λόβιν, και εγώ θα ήθελα να μάθω τις πρόσφατες εκτιμήσεις, τις τελευ... τα τελευταία στοιχεία για την κατάσταση των κεφαλόποδων. Επίσης ε, έγινε μια αξιολόγηση του αντικτύπου της υποχρέωσης εκφόρτωσης, γιατί θέλουμε πραγματικά μια επικερδή αποφελή συμφωνία για όλα τα συμβαλόμενα μέρη, και τους Μαυριτανούς και τους Ευρωπαίους, για να μπορούν και οι δύο πλευρές να βγουν κερδισμένες και να περιοριστεί όσο γίνεται ο κοινωνικός αντίκτυπος. Ευχαριστώ κύριε Μιράντα. Ευχαριστώ. Και εγώ κατάγομαι από, μια, από ένα έθνος ελευθερικό από τα πιο σημαντικά της Ευρώπης που εξαρτάται πλήρως από την Αλία και κυρίως από την παράκτη Αλία. Γι' αυτό και θα ήθελα να πω ότι σεβόμαστε πλήρως τους εκπροσώπους ε, και της πελαϊκής αλίας και της παράκτης αλίας μικρής κλίμακας αλλά είμαστε υπέρ και της ε, ε, αλληλευτική και κυριαρχίας της Μαυριτανίας. Είμαστε μια χώρα, όπως είπα, που εξαρτάται από την αλία χταποδιού. Το χταπόδι αποτελεί τμήμα του πολιτισμού μας, της κουλτούρας μας. Έχει λοιπόν και πολιτιστική διάσταση και αλληλευτική διάσταση και προσαρμόζουμε πολλά αλληλευτικά σκάφη στην αλία χταποδιού. Έχω λοιπόν μια ερώτηση στους ε, δύο εμπειρογνώμονές μας αναφέρθηκε περιλημμένως η κατάσταση του αποθέματος χταποδιού. Γιατί πιστεύετε ότι η Μαυριτανία έκανε υποχωρήσεις ε, σε άλλες χώρες. Γιατί για υποχωρήσεις ε, μιλάμε. Όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε άλλες χώρες. Γιατί λοιπόν ενώ αρνηθήκατε αυτή την πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνατε, επιτρέψατε σε άλλε χώρε να λιεύσουν κεφαλόποδα, αν υποτίθεται ότι το χταπόδι βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Από ό,τι φαίνεται, τελικά δεν βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Νομίζω ότι είναι κάπω αντιφατική αυτή η στάση τη Μαυριτανία. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε τι ερωτήσει. Θα περάσουμε τώρα στο γύρο των απαντήσεων. Παρακαλώ να είστε όσο πιο συνοπτικοί γίνεται και συγκεκριμένοι για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ποιο εμπειρογνώμονα θέλει το λόγο για να απαντήσει. Ο κύριος Καγιάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει λοιπόν το θέμα της κατάστασης από θέματος χταποδιού. Εγώ αναφέρθηκα σε μελέτες του 2009 και του 2010 που έγιναν σε διεθνές επίπεδο. Η ΚΟΠΑΣ ε, οργάνωσε της ΦΑΟ ανέθεσε σε ξένους εμπειρογνώμονες στην ε, κατάρτιση αυτών των μελετών. Δεν ξέρω τι είπε το Ισπανικό Καιρογραφικό Ινστιτούτο για την κατάσταση αυτή με πιο πρόσφατα στοιχεία. Πάντως η ΕΤΟΕΑ, η Ευρωπαϊκή ε, Κοινωνική και Επιστημονική Επιτροπή, ουσιαστικά ενέκρινε μία εναλλακτική μέθοδο διαχείρισης για να, να βελτιωθεί η διαχείριση του χταποδιού προσδιορίζοντα διαφορετικά τι ζώνε, ανοίγοντα και κλείνοντα μερικέ ζώνε. Δεν ήταν όμω μια διαδικασία αξιολόγηση του αποθέματο. Τώρα, αν θα πρέπει να γίνει με βάση τα νέα στοιχεία κάτι για τη συμφωνία, κατά τη γνώμη μου ίσως θα πρέπει να συνεδριάσει πρώτα η μεικτή επιστημονική επιτροπή. Πρόκειται για ένα όργανο που δημιουργείται από τη συμφωνία, νομίζω ότι αυτή η μεικτή επιτροπή είναι κατάλληλη και αρμόδια να κάνει μια ανεξάρτητη αξιολόγηση. Να δούμε τα στοιχεία και όχι μόνο τις μελέτες. Γιατί αυτό είναι νομίζω το πρώτο απαραίτητο στάδιο. Δεύτερον, κύριε Λόβιν, ρωτήσατε για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της συμφωνίας. Και του Ευρωπαϊκού Ελευτικού Στόλου, αλλά και γενικώ των ελευτικών στόλων. Ο Ευρωπαϊκός Ελευτικό Στόλος, όπως και, και ο στόλος της Μαυριτανία, ε, χρησιμοποιούν μηχανότρατες κυρίως. Οι μηχανότρατες, ξέρετε, έχουν κάποιο περιβαλλοντικό αντίκτυπο, γιατί επηρεάζουν ε, το βυθό, Παλιεύουν στο βυθό και άρα αγγίζουν πολλά αλλιευτικά είδη. Οπότε υπάρχει περιβαλλοντικός αντίκτυπος. Αλλά ο ίδιο είναι και για τα μαυριτανικά σκάφη και για τα ευρωπαϊκά. Έχουμε 100 σκάφη της Μαυριτανία για τα κεφαλόποδα, ενώ 30 είναι τα ευρωπαϊκά αλληλευτικά σκάφη που αλληλεύουν κεφαλόποδα. Ίσως υπάρξουν κάποιες λύσεις, θα πρέπει να τις αναζητήσουμε και εκεί θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στη μελλοντική συνεργασία. Δηλαδή, αναζήτηση της επιλεκτικότητας, που ήταν μέχρι στιγμής ο φτωχός συγγενής της αλληλευτικής σύμπραξης. Κακός. Γιατί αν δώσουμε την έφταση στην επιλεκτικότητα των τρατών, με βάση τη δική μας την ευρωπαϊκή εμπειρία, θα μπορούσαμε να μειώσουμε, να περιορίσουμε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Γιατί αυτός ο αντίκτυπος είναι ούτε χειρότερος ούτε χαμηλότερος από τον ένα στο όλο στον άλλο. Απλώς θα πρέπει να τον μετριάσουμε με κάποιο τρόπο. Αυτά ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τον κύριο Βουλευτή και την κυρία Βουλευτίνα ότι στη Μαυριτανία το χταπόδι είναι στατηγικό αλίευμα για τη Μαυριτανία. Και μόνο οι Μαυριτανοί το αλλιεύουν, κανένας ξένος. Δεν έχει την άδεια να ψαρέψει χταπόδι. 36.000 ε, αλληλείς είναι Μαυριτανοί όλοι που ασχολούνται με το χταπόδι. Κανένας μη Μαυριτανός δεν μπορεί ούτε κάποιος από τη Γκάμπια ούτε τη Σενεγάλη να μπορεί να εκφορτώσει αυτό το λίγο. Ζητώ να έρθουν στο Νιομπού να δουν τι γίνεται στις εκφορτώσεις επιτόπου. Λοιπόν, και γίνεται, ε, γίνεται και έλεγχος όσον αφορά τη μεταφόρτωση. Κανένας ξένος δεν αλλιεύει το χταπόδι. στρατηγική σημασία και τη Μαυριτανία. Στο Υπουργείο Αλλιές υπάρχει μία άδεια πελαγική και για τα άλλα είδη και ξεχωριστή για το χταπόδι. Δεν υπάρχει κανένας ξένος αλλοδαπός στον τομέα του χταποδιού. Δεν επιτρέπεται κανείς άλλος να αλλιεύσει στη Μαυριτανία και ούτε στους Κινέζους το επιτρέπουμε. Μόνο με τα πελαγικά είδη ασχολούνται. Εμείς ήμασταν κατά αυτής της συμφωνίας. Είμαστε κατά ε, οποιοδήποτε ξένου που θα μπορούσε να λιεύσει ένα, ε, ένα, και ένα χταπόδι. Για τα πελαγικά είδη υπάρχουν ένα 1.200.000 τόνοι που μπορούν να ληφθούν στα πελαγικά. 300 πυρούγες ε, επιτρεπόταν ε, από τους Σενεγαλές να λιεύουν. Ε, και υπάρχουν ναυλωμένα πλοία που ασχολούνται με τα πλαγικά. Στον τομέα του χταποδιού κανένα ξένο καράβι δεν μπορεί να ψαρέψει χταπόδι στη Μαυρτανία. Το δεύτερο πρόβλημα. Λοιπόν, ετοίμασε πρόγραμμα χρηματοδότησης εργαζομένων στα ευρωπαϊκά σκάφη και ε, έχουν τα δικά του σκάφη και εργάζονται, αυτοί που εργαζόταν στα ευρωπαϊκά πλοία εργάζονται στον τομέα του χταποδιού. Και για, τα, για την πελογική αλία ε, οι ναυτικοί πήγανε στα πλοία αυτά. Δεν τίθεται πρόβλημα στη Μαυριτανία. Θα υπάρξει και χρηματοδότηση. Η βιοτεχνική αλία είναι ανάπτυξη. Για 10.000 ευρώ μπορείτε να δημιουργήσετε 12 θέσεις απασχόληση. Όσον αφορά το χταπόδι, τα αποθέματα χταποδιού, έχουμε Ινστιτούτο και Αναγραφικής έρευνα Αλία στη Μαυριτανία που κάνει αξιολογήσει κάθε τέσσερα χρόνια. Και όλοι οι εμπειρογνώμονε οι Ευρωπαίοι παρέσταν στην τελευταία αξιολόγηση του 2010. Έγινε παρουσία των πάντων. Εμεί οι επαγγελματίε ήμασταν παρόντε είχαμε πρόσβαση, μπορέσαμε να παραστούμε στην αξιολόγηση. Το ξέρουν οι αλείς. Πάνω 50.000 τόνους στην καλύτερη χρονιά στο χταπόδι δεν μπορούμε να φτάσουμε. Σήμερα είμαστε στους 27.000 τόνους. Υπάρχει υπερεκμετάλλευση. Του ΙΜΡΟΠ στις εκθέσεις είδαμε ότι πρέπει να μειωθεί κατά 5%, 40%. Έγιναν συλλήψεις. Εμείς την περίοδο ε, Μαΐου-Ιουνίου, Σεπτεμβρίου σταματούμε την περίοδο της πάυσης. Είναι περίοδος αναπαραγωγής. Αναπαράγεται κυρίως αληφτικές ζώνες το χταπόδι και σταματάμε. Και τηρούμε αυτή ε, την περίοδο της γεννήσεων και ανάπτυξης του χταποδιού. Και στο ΙΜΡΟΠ γίνονται επαφές μεταξύ επαγγελματιών και επιστημόνων πάνω σε αυτό. Κάνουμε μια παύση το προτείνουμε στι αρχές. Αυτό γίνεται και είναι σωστή διαχείριση. Κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες η Μαυριτανία για διατήρηση ε, του θαλασσίου περιβάλλοντος. Γι' αυτό το χταπόδι αρχίζει να σώζεται. Κάποια περίοδο ούτε δύο τόνους την ημέρα χταπόδι δεν ψαρεύαμε κάποια περίοδο. Σήμερα που ξανάρχισε η περίοδος είμαστε στους 150 τόνους την ημέρα στο Μαλιμπού και μειωθήκαμε τώρα στους 30. Και λέει η μελέτη ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση ε, το χταπόδι. Οι αλλοίς γνωρίζουν ότι υπήρχε αυτό και υπάρχει ένα πρόγραμμα διαχείρισης που εφαρμόζεται. Μέχρι 70 χιλιοστά το μάτι του δικτύου μεγαλώσαμε. Ε, κλείνουμε διάφορες ζώνες το ζητά ο τομέα. Θέλουμε να διατηρηθεί το χταπόδι, να το προστατεύσουμε το χταπόδι. Το χταπόδι είναι αυτό που μας βγάζει, με το οποίο βγάζουμε το ψωμί μας. Ε, δεν αρκεί έτσι. Δεν μπορούμε να βρούμε κάτι άλλο. Για τα πελαγικά, κάντε επενδύσει στα πελαγικά. Γιατί δεν είδαμε εργοστάσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ βλέπουμε κινέζικα εργοστάσια. Κάντε εργοστάσια. Κάντε να εργαστούν τα πλοία σα ε, εκφορτώστε, δώστε προστιθέμενη αξία. Εμείς δεν κερδίζουμε τίποτα τα σκάφη. Χρειάζεται ανάπτυξη. Αυτό είναι σημαντικό. Να εργάζεται ο πληθυσμός. Να κερδίζει κάτι από τι σημαντικέ συμφωνίε. Εάν δεν υπάρχει αυτός αντίκτυπος, εάν δεν προστίθεται αξία για τον πληθυσμό. Αν δεν έχει αξία ο πληθυσμό, όπω προανέφερα κάποια χρόνια πριν, κάντε να συμμετέχει ο κόσμο, ο ντόπιο πληθυσμό, οδηγήστε στην ανάπτυξη, μιλήστε εργοστάσια, να είσαστε πιο κοντινοί με εμά. Συνεννοούμαστε, κάντε κάτι. Να υπάρχει σωστή συνεργασία, δίκαιη συνεργασία, αναπτυξιακή συνεργασία. Αυτό είναι σημαντικό. Αν είναι να έρχεστε να ψαρεύετε και να φεύγετε, τι να κάνουμε. Εμεί παίρνουμε 50% από τα πελαγικά σκάφη τα πελαγικά σκάφη παίρνουν από την στροφά μας και την τσιπούρα μας. Λοιπόν, 50% τσιπούρας μας παίρνουμε. Ε, το βλέπετε εδώ. Για να σας πω ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε πραγματική εταιρική σχέση, ε, διαφανή. Θέλουμε να αλλιεύετε εσείς και εμείς να αναπτυχθούμε. Αυτό είναι σημαντικό. Εάν δεν γίνει αυτό, δεν ξέρω τι να πω. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά ξεπεράσετε πολύ την εμβέλεια των ερωτήσεων και δεν έχουμε και χρόνο στη διάθεση μας. Ευχαριστούμε πάντως για τις απαντήσεις. Ο κύριος Γκαράτ. Ευχαριστώ. Και εγώ συμφωνώ με τις τελευταίες παρατηρήσεις του εκπροσώπου του Μαυρετανικού Ελευτικού Στόλου. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω η κατάσταση αυτή να θεωρηθεί ως ε, ε, πόλεμος μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ελευτικού Στόλου και του Μαυριτανικού. Και εμείς ε, ε, θέλουμε να προστατευτεί, να διαφυλαχθεί η παράκτη αλία της Μαυριτανίας και ο τοπικός στόλος και τους ευχόμαστε καλή τύχη. Και όπως είπατε, η ευρωπαϊκή αντιπαροχή δεν θεωρήθηκε πολύ σημαντική για, για τους τοπικούς ψαράδες, σε αντίθεση με τις αντίστοιχες επενδύσεις των ε, Κινέζων, των ε, Ιαπώνων, που είχαν πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια και φαίνονται παντού αφήσει με ευχαριστίες προς τους Κινέζους και τους ε, Ιάπωνες, ενώ η ευρωπαϊκή συρισφορά ήταν ελάχιστη και δεν έγινε καθόλου αισθητή σχεδόν από τοπικό πληθυσμό. Κύρια Λόβιν, για τις δύο μελέτες του Ισπανικού Οκεανογραφικού Ινστιτούτου. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια διαφοροποίηση μεταξύ της κατάστασης του κεφαλοπόδου και των χταποδιών αφενός και του θέματος των πλεονασμάτων και αν θα πρέπει να αλλιεύουν τα πλεονάσματα οι Ευρωπαίοι. Σε ό,τι αφορά την πρώτη μελέτη του Ισπανικού Οκεανογραφικού Στούτου, εκεί αναφερόταν ένα μοντέλο ε, τοπικής, ε, τοπικού αποκλεισμού, χωρικού αποκλεισμού, όχι μόνο για, για τον Ευρωπαϊκό Στόλο, αλλά και για, την, για το στόλο της παράκτης ελίας μικρής κλίμακας της Μαυριτανίας και μάλιστα υπευλήθη αυτό στην κοινή επιστημονική επιτροπή, στη μεικτή επιστημονική επιτροπή και εκεί ακούστηκε ότι αν λεφθούν κάποια μέτρα διαχείριση για απαγόρευση της αλίας σε συγκεκριμένες περιόδους του χρόνου, σε συγκεκριμένες εποχές και για τους δύο στόλους θα μπορούσαμε να έχουμε ε, δυναμικό παραγωγής ε, αχταπόδιου πάνω από 60.000 τόνους, δηλαδή το διπλάσιο από ό,τι αλλιεύεται σήμερα. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Αυτό που εμείς ενθαρρύνουμε τις μαυρετανικές αρχές να κάνουν και την παράκτεια μικρής κλίμακας ελίας είναι να εφαρμόσουν αυτό το μοντέλο ε, χωρικού αποκλεισμού, γιατί θα αυξηθεί η παραγωγή. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αυξηθεί η δυνατότητα παραγωγής, που είχε μειωθεί τον τελευταίο καιρό. Επίσης, να υπενθυμίσω ότι τα μικρά ελευτικά σκάφη δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ε, ε δίκτυα άνω των δύο μέτρων και υπάρχει η ασυμβατότητα με την απαγόρευση στα 6 μίλια. Τώρα μιλάμε για 60.000 τόνους ε, δυναμικό. Εμείς αρκούμαστε και στις 6.000 τόνους που είναι ελάχιστη ποσότητα σε σχέση με το δυναμικό παραγωγής και είμαστε επιπισμένοι ότι μπορούμε κάλλιστα να συνεπάρξουμε με το μαυριτανικό αλληλευτικό στόλο γιατί ο η παράκτη λία τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έδρα τη Κανάρια νησιά και τη Γαλλικία κυρίω. Τώρα, μετά τι παρατηρήσει που κάναμε, τη δειγματοληψία και τα στοιχεία από τα αλεύματα, έχουμε ε, τη μελέτη του 2012 του Οκεανογραφικού Ινστιτούτου. Εκεί, εκεί φαίνεται μια πολύ καλή κατάσταση του αποθέματος του χταπόδιου και μάλιστα υπάρχει μια θετική τάση και ανωδική Βλέπετε εδώ ότι την τελευταία χρονιά, βλέπετε στον πίνακά μου, είχαμε την τελευταία χρονιά μια σημαντική αύξηση των αλλιευμάτων, της αλλιεύσης του χταποδιού. Όχι ότι έχει αυξηθεί ο τρόπος ε, διαχείρισης, αλλά έχει, αυξηθεί η παρουσία του χταποδιού, γι' αυτό και αλλιεύεται πολύ περισσότερο χταπόδι. Τώρα, για να λυθούν οι αμφιβολίες και οι απορίες, γιατί άλλο λέει ένας και άλλο λέει άλλος, θα έλεγαμε η Μικτή Επιστημονική Επιτροπή με εμπειρογνώμονες και των δύο πλευρών να συνέλθει το συντομότερο δυνατό και να εκφέρει τη γνώμη της για το ποια είναι η κατάσταση του χταποδιού. Τώρα, άλλο αν η κυβέρνηση Μαυριτανίας θέλει το θεωρητικό πλεόνασμα που θα δημιουργηθεί να το αλλιεύουν οι Ευρωπαίοι ή άλλοι. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Θα σεβαστούμε την απόφαση τη Μαυριτανική κυβέρνηση. Αυτό που λέμε είναι ότι αν υπάρχει πλεόνασμα, αν διαπιστωθεί, να το αλλιεύσουμε εμεί. Μα ενδιαφέρει. Αλλιώ θα το κάνουν οι Κινέζοι. Αυτή τη στιγμή κανένα κινέζικο σκάφο δεν αλλιεύει στην περιοχή, αλλά μέχρι πρόσφατα ήταν πέντε τα σκάφη της, τα κινέζικα που αλλιεύαν κεφαλόποδα. Τώρα για τη δεύτερη ερώτηση. Τι κάνουμε τώρα. Νέα διαπραγμάτευση ή μπορεί να γίνει κάποια διόρθωση του υφιστάμενου πρωτοκόλου. Εμείς θα προτιμούσαμε το συντομότερο δυνατό να ξανακάτσουν στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Μαυρετανία και να εξετάσουν την κατάσταση γιατί δεν ψαρεύουν οι Ελλείς παρά την αλληλευτική συμφωνία. Ποια τεχνικά προβλήματα υπάρχουν και να υποβάλουν μια καλύτερη πρόταση. Αν δεν γίνεται δυνατό κάτι τέτοιο από νομική άποψη, τότε το μόνο που μένει είναι να καταγγελθεί η συγκεκριμένη συμφωνία και να γίνει διαπραγμάτευση μια νέα συμφωνία. Γιατί όλο και αν επιμένω να το προσπαθήσουμε, αν μια επιχείρηση ξέρει ότι θα στείλει σε, σε ζημία σίγουρη το σκάφος δεν πρόκειται να το στείλει. Αυτό συμβαίνει και για τα πελαγικά είδη και για τα θαλασσινά. Ε, τα σκάφη που αλληλεύουν κεφαλόποδα είναι δεμένα στα λιμάνια. Και οι βοήθειες, ε, οι ενισχύσεις θα σταματήσουν. Οπότε θα απολυθούν οι ναυτικοί και θα μείνουν στα λιμάνια τα πλοία. Αυτό είναι κρίμα και για την Μαριτανία αλλά και για τη Γαλλικία και τα Κανάρια νησιά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βαμπάλσορ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σύντομα. Δεν υπήρξαν ε, ερωτήματα προς, σε σχέση με αυτά που είπα, άρα είναι σαφή. Θα ήθελα μόνο να σχολιάσω αυτά που είπε ο συνάδελφος από τη Μαυριτανία. Μίλησε για τα παραλιεύματα, τα κεφαλόποδα παραλιεύματα. Πάντα παρατηρούσαμε βεβαίω τι ε, μηχανότρατε που αλλιεύουν στην ε, Μαυριτανία και δεν είχαμε παρατηρήσει ότι υπήρχαν κεφαλόποδα ω ε, παραλλιεύματα. Ήθελα απλώ να το καταστήσω σαφέ. Δεν ξέρω αν εννοούσε αυτό ο κύριο από την Μαυριτανία. Εγώ έτσι το κατάλαβα. Δεν έχουμε κεφαλόποδα στην πελαγική αλλιεύμα μα ω παραλλιεύματα. Καλώ. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση και ευχαριστώ τους εμπειρογνώμονές μας για τα πολύ διαφωτιστικά του σχόλια. Τους ευχαριστώ και πάλι θερμά και έχουμε 25 ακόμη λεπτά για τη δεύτερη ενότητα, το δεύτερο τμήμα της συζήτησης που αφορά την εξέταση της δικής μου έκθεσης. Και μια και εγώ είμαι ο εισηγητής εδώ, θα ήθελα να δώσω την προεδρία στον συνάδελφο για να κάνω εγώ την παρουσίαση. Okay. Uh, I hope I won't uh, make the same mistakes according to according to names as last time. Την προηγούμενη φορά προσπάθησα να αυτοπεριοριστώ κι εγώ, αλλά και να περιορίσω και εσάς ε, που θα συμμετέχετε στη συζήτηση. Θα ξεκινήσουμε δίνοντας το λόγο στον εισηγητή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήδη είναι δεύτερη τρίτη φορά που εξετάζουμε αυτό το θέμα. Ήδη είχαμε εκτενείς συζητήσεις και πολύ καλές και μάλιστα και σήμερα είχαμε πολύ χρήσιμη ακρόαση για αυτό το σημαντικό αυτό θέμα. Θα είμαι λοιπόν λακωνικός και θα περιοριστώ σε τρία σημεία που κατά τη γνώμη μου είναι κέρια και συνοψίζουν κάλλιστα την έκθεσή μου. Λέω καταρχήν ρητά και κατηγορηματικά εγώ ότι είμαι υπέρ μια αλληλευτική συμφωνία με τη Μαυριτανία. Γιατί θεωρώ ότι μια τέτοια απόφαση είναι υποφελή και για τη Μαυριτανία και για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν θέλω τη συγκεκριμένη συμφωνία, γιατί αυτή η συγκεκριμένη συμφωνία δεν είναι καλή. Είναι κακή, όπω φάνηκε ξεκάθαρα. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε τη σημαντικότερη ε, αλληλευτική συμφωνία σε ό,τι αφορά τον όγκο, την ποικιλία των αλληλευτικών ε, ειδών, αλλά και τη μεγαλύτερη χρηματική αντιπαροχή. 70 εκατομμύρια ευρώ και επιπλέον το χρηματοπιστωτικό αντιστάθμισμα που θα δώσει ο τομέα με τη μορφή κανόνα. Βέβαια, παρόλα αυτά, ο κλάδο μα δεν χρησιμοποιεί τι αλληλευτικές δυνατότητε που έχει. Γιατί? Γιατί υπάρχει πρόβλημα. Θα πρέπει, αν μη τι άλλο, να καθίσουμε και να σκεφτούμε το θέμα και να δούμε γιατί οι αλληλείς που είναι οι δικαιοχευτές συμφωνίας ε, την απορρίπτουν. Κάπου υπάρχει πρόβλημα. Και φτάνω εδώ στο δεύτερο σημείο, που είναι πολύ σημαντικό. Ας μην ξεχνούμε ότι έχουμε μία αλλιευτική συμφωνία εδώ. Επαναλαμβάνω, η συμφωνία είναι αλλιευτική. Και το θέμα είναι πολύ σημαντικό, το ξεχνάμε μερικές φορές. Ακόμη και σήμερα φάνηκε από μερικές περιπτώσεις ότι το ξεχνάμε αυτό. Είμαστε αλληλευτική επιτροπή και εξετάζουμε μία ε, συμφωνία αλληλευτικής σύμβασης και τα συναφή πρωτόκολλα, που είναι α, κυρίως εμπορικά, αφορούν την αλία και δεν πρόκειται για συμφωνίες αναπτυξιακή συνεργασία ή άλλου είδου συμφωνίε. Είναι αλλιευτικέ εμπορικέ συμφωνίε μα, κατά κανόνα. Άλλωστε, με βάση τη συνθήκη, έχουμε την εντολή να έχουμε ε, και τέτοιες αναπτυξιακές συμφωνίες. Είναι το άρθρο 208 της, ε, συμφωνίας, της ε, Συνθήκη Λισαβόνα, αυτή η νομική βάση, αλλά η δική μας νομική βάση είναι το άρθρο 218 που αφορά τι ελευτικές συμφωνίε. Μην ξεχνάμε λοιπόν και τη νομική βάση. Λοιπόν, πρόκειται για μια αλληλευτική συμφωνία που με βάση κάποιο χρηματοοικονομικό αντιστάθμισμα λαμβάνει χ αλληλευτικέ δυνατότητε. Και με βάση αυτό το στοιχείο θα πρέπει να καταλήξουμε στο χαρακτηρισμό τη συμφωνία ω καλή ή κακή. Άσχετα με τα υπόλοιπα θέματα που δεν αφορούν την αλληλεία. Βέβαια, η συμφωνία και τη αλληλευτική έχει κάποιες επιδράσεις και σε άλλα θέματα. Έχουμε 3 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα από την περασμένη φορά. Γιατί δεν είχαν εγκριθεί τόσο σημαντικά ποσά. Και τώρα, από αναπτυξιακή άποψη, αρμόδια είναι η Επιτροπή ΔΕΒΗ, η Επιτροπή Ανάπτυξης. Εκεί θα δώσει μια διαφορετική ανάλυση της κατάστασης υπό το πρίσμα της ανάπτυξης. Εμείς δίνουμε την ανάλυση μας υπό το πρίσμα της αλίας. Επαναλαμβάνω, η συγκεκριμένη συμφωνία και το συγκεκριμένο πρωτόκολλο είναι επιζήμια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά είναι αρνητική ακόμη και για τη Μαυριτανία, μια που δεν ε, αλλιεύει ο στόλος. Δεν πρόκειται να εμβαθύνω σε όλα τα σημεία γιατί τα είδαμε. Βλέπετε και στην έκθεση ότι αμφισβητώ και την ίδια δυναμική βάση. Είναι ένα άλλο ακόμη θέμα ε, τυπικό περισσότερο, αλλά είναι περίεργο που το Συμβούλιο άλλαξε την νομική βάση και απέριψε, ε, εξάλληψε την παραπομπή στο 43.2. Έμεινε μόνο η παραπομπή στο άρθρο 43, χωρίς να φέρει το εδάφιο 2. Ένας λόγος λοιπόν παραπάνω για να πούμε ότι δεν μας αρέσει αυτή η προσέγγιση του Συμβουλίου για το θέμα αυτό. Εγώ τώρα θα επικεντρωθώ σε δύο βασικά σημεία. Η συμφωνία ε, δίνει μικρότερες αλληλευτικές δυνατότητες από την προηγούμενη και μάλιστα σε χειρότερες συνθήκες. Επιπλέον η συμφωνία είναι εξαιρετικά δαπανηρή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και βλέπουμε και από τον τομέα ότι οι άδειες αυξάνονται. Μιλάμε για ποσοστό που αφισβητείται, αλλά είναι πολύ υψηλότερο από ό,τι οι ελευτικές δυνατότητες. Τώρα, για τα κεφαλόποδα. Η κατάσταση είναι φως φανάρι. Δεν υπάρχει πρόσβαση καν στο αλληλευτικό αυτό είδος, παρόλο που προβλέπεται αναθεώρηση μετά από ένα χρόνο. Η αναθεώρηση αυτή είναι απαραίτητη, γιατί εμείς ε, αμφισβητούμε ε, την ε, αναθεώρηση μετά από ένα χρόνο. Γιατί σε μια εμπορική συμφωνία που η διαπραγμάτευσή τη κράτησε 15 μήνε και η ισχύ τη θα είναι διετή, θα πρέπει από τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει να διαπραγματεύεται την, την αναθεώρηση τη συμφωνία. Αλλιώ θα περάσουν πολύ γρήγορα τα χρόνια. Η αναθεώρηση είναι απαραίτητο να γίνει μετά από ένα χρόνο όταν η χρηματική αντιπαροχή έχει ήδη δοθεί 70 εκατομμύρια ευρώ που προς τίθεται στη δυνατότητα αλίας και κεφαλόποδων. Ενώ φαντάζομαι ότι αν προσταθούν τα κεφαλόποδα η Βαβριτανία θα ζητήσει επιπλέον χρηματικό αντιστάθμισμα. Κάτι που δεν πιστεύω ότι θα γίνει, οπότε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. 32 σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μείνουν χωρίς αλληλευτική ζώνη και χωρίς εναλλακτική λύση. Το πιο σημαντικό είναι πάντως και φάνηκε εδώ, είναι ότι η απαγόρευση αυτή ε, τεκμηριώθηκε με βάση παροχημένα επιστημονικά στοιχεία. Μας το είπε εμπειρογνώμονας. Επρόκειτο για στοιχεία του 2008, του 2009, παροχημένα. Δεν υπάρχουν επίκαιρα στοιχεία που να τεκμηριώνουν αυτή την, από, την, τον αποκλεισμό. Το αντίθετο. Σήμερα, με βάση τις νέες επιστημονικές μελέτες, το επίπεδο των κεφαλόποδων όχι μόνο δεν είναι κακό, αλλά είναι μάλλον σε επίπεδο μέγιστης βιώσιμης απόδοσης. Υπάρχει με βελτίωση έως και 30% σχέση με το παρελθόν. Οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε για υπερεκμετάλλευση του χταποδιού, όπως ε, έλεγε το παλιό μας ψήφισμα. Σήμερα μια τέτοια διαπίστωση είναι ανεδαφική, παροχημένη. Γιατί εμείς καταρχήν ήμασταν υπέρ του αποκλεισμού των κεφαλοπόδων εξαιτία τη υπερεκμετάλλευση που είχαμε διαπιστώσει, αλλά στο μεταξύ έχουν αλλάξει τα επιστημονικά στοιχεία. Δεν υπάρχει πια υπερεκμετάλλευση. Το αντίθετο. Οι αρχές της Μαυριτανίας θέλουν ε, το πλεόνισμα να το κρατήσουν για τους δικούς τους ελίους, τους ντόπιου. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε προσαρμογή της συμφωνίας στα νέα στοιχεία, στην πραγματικότητα. Και συμφωνώ ότι και ο στόλος Μαυριτανίας θα πρέπει να έχει πρόσβαση στους πόρους, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν αρκετοί πόροι για την εκμετάλλευση της βιομάζας του χταποδιού και για τους δύο στόλους. Σε ό,τι αφορά τα πελαγικά είδη, εκεί φάνηκε ότι η μετατόπιση της αλληλευτικής ζώνης ε, γίνεται χωρίς αύξηση των αλληλευτικών δυνατοτήτων. Κάτι που σε τελική ανάλυση μας εκπλήσει. και δημιουργεί ένα επιπλέον ερωτηματικό, όπως η υποχρεωτική εκφόρτωση στη Μαυριτανία, η υποχρεωτική μεταφόρτωση, κάτι που αφισβητήθηκε και από τον τοπικό πληθυσμό. Όλα αυτά φέρνουν σε δύσκολη θέση τον ελευτικό στόλο και θα ήθελα να κάνω και μία σύντομη αναφορά στα Κανάρια νησιά, για προφανείς λόγους ευνόητους, την υποχρέωση εκφόρτωση στη Μαυριτανία. Αυτό θα είναι πολύ αρνητικό για την οικονομία και την απασχόληση μιας περιφέρειας Ευρωπαϊκής Ένωση που έχει ποσοστά ανεργία πάνω από 36%. Μιλάμε για 2.750 θέσει εργασία άμεσα συνδεόμενες με την Αγγλία και με δραστηριότητα λιμενική περίπου 40 εκατομμυρίων. 300 ε, εκατομμυρίων. Άλλωστε η Ευρωπαϊκή Ένωση που επένδυσε σε επενδύσεις, ε, που επένδυσε σε υποδομές τεράστια κονδύλια στη, στη Πάλμας. η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση που χρηματοδότησε αυτές ε, τις υποδομές να τις οδηγήσει σε καταστροφή, γιατί σε αυτό θα καταλήξουμε αν εγκαταληφθούν οι δραστηριότητες, σε ό,τι αφορά τα βεθοπελαγικά και τα θαλασσινά. Το ίδιο δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε. Για μία ακόμη φορά η, η μετατόπιση των ελευτικών ζωνών δημιουργεί τεράστια απώλεια αποδοτικότητα στον κλάδο. Γιατί στις παλιές ζώνες ε, είχαμε μεγάλη συγκέντρωση της αλίας καραβίδας κυρίως. Τώρα, για μία ακόμη φορά μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν εύλογοι λόγοι ή τεκμηριωμένα επιστημονικά πορίσματα που να στοιχειοθετούν ε, ή να δικαιολογούν μάλλον τη μετατόπιση των ελευτικών ζωνών. Και ένα άλλο θέμα είναι το υπέροχο ποσό της χρηματικής ε, αντιπαροχής που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 110 εκατομμύρια ευρώ περίπου, πολύ δαπανηρή συμφωνία. Από αυτά 77 είναι για τους πόρους 40 ε, είναι ε, η προσπάθεια του τομέα. Είναι πολύ δαπανηρή λοιπόν αυτή η αλληλευτική συμφωνία. Θα μπορούσαμε να την αναλάβουμε αυτή την αντιστάθμιση αν είχαμε μία αντίστοιχη παροχή από την Μαυριτανία με τη μορφή ελευτικών αδεών και προϋποθέσεων που θα ήταν αποδεκτές από το δικό μας ελευτικό στόλο. Κάτι που είναι σημαντικό για την έκθεση και τη συμφωνία είναι ποια είναι η θέση των δικαιούχων. Γιατί ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Είναι η κοινωνία της Μαυριτανίας και ο αλληλευτικός στόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη ο αλληλευτικός, οι αλληλείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης είπαν όχι στη συμφωνία. Και θα πρέπει να μας το εξηγήσει επιτέλους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί από την πρώτη στιγμή δέχτηκε μία αντιπαροχή 70 εκατομμυρίων ευρώ, την ίδια δηλαδή που είχε μέχρι τώρα, παρόλο που έχουν αφαιρεθεί τα, χτα, τα, κεφαλόποδα, το, το χταπόδι. Γιατί, ενώ αφαιρέθηκε ένα είδος, ε, έμεινε ίδιο το ύψος της αντιπαροχής. Εγώ συμφωνώ με το δικαίωμα να αλλιεύουν οι Μαυριτανοί το χταπόδι, αλλά γιατί να μην μειωθεί ε, το αντίστοιχο αντιστάθμισμα εφόσον έχουμε αποκλειστεί από το χταπόδι. Αυτά. Επίσης έχω ευξηθεί το κόστος των αλλιευτικών αδειών. Επαναλαμβάνω, δεν είναι επικερδής η συμφωνία, δεν είναι κερδοφόρη η η χρήση των αλλιευτικών δυνατοτήτων είναι κοντά στο μηδέν ο κλάδος τον απορρίπτει και μάλιστα και πριν τη διεκπαιρέωση των διαπραγματεύσεων το είχε επισημάνει αυτό ο κλάδος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την είναι κακή συμφωνία και παρόλα αυτά η Επιτροπή τον αγνόησε. Αυτά. Επαναλαμβάνω. Ήταν πολύ χρήσιμη και ενδιαφέρουσα η σημερινή ακρόαση. Και μετά από αυτήν όχι μόνο επιμένω στην ε, διαφωνία μου με, τη με την ε, ληφτική σύμπραξη, αλλά και θεωρώ ότι είναι άσκοπο να επιμένουμε σε μια κακή συμφωνία, που είναι κακή όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τη Μαυριτανία. Ευχαριστώ κύριε Ματοντροβέρ. Τέθησαν πολλές ερωτήσεις που απευθυνόταν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να πάρει το λόγο σε αυτό το στάδιο ή να μπούμε στη συζήτηση. Ο κ. Σάντσες αντί αυτή την περίπτωση έχει το λόγο. Eh, mm, Ευχαριστώ. Δεν θα επαναλάβω αυτά που ακούσαμε από τον εισηγητή μας, τον κύριο Μάτο. Θα ήθελα απλώς να επαναλάβω ότι πολύ θα ήθελα να πονέσει την στην αυτή συμφωνία με τη Βρετανία, αλλά δυστυχώ έχω πολύ σοβαρέ ακόμη επιφυλάξει και ενδιασμού. Εγώ είμαι υπέρ τη αναδιαπραγμάτευση. Γιατί άλλο είναι αναπτυξιακή ε, βοήθεια και άλλο η αλληλευτική συμφωνία. Γιατί η αναπτυξιακή συμφωνία δεν συνοδεύεται από χρηματικό αντιστάθμισμα, από αντιπαροχή. Εκεί θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συνεργασία με τη Μαυριτανία. Ανεπιφύλακτα και ανεφόρον και θέλουμε να αξιοποιηθεί. Αλλά όταν έχουμε μια αλληλευτική συμφωνία, χρειάζεται κάτι επιπλέον, χρειάζεται μια αντιπαροχή. Και φυσικά χρειαζόμαστε απόλυτη διαφάνεια και ισορροπία μεταξύ της βιωσιμότητας αλίας και της συμβολής στην βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια, είναι προφανές ότι σήμερα διασκεδάστηκαν κάποιες ανησυχίες, αλλά υπάρχουν αμφιβολίες και για την κατάσταση των αποθεμάτων, αλλά υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν συναυθεί διμερείς ιδιωτικές συμφωνίες με τις μαυρετανικές αρχές. Οπότε μπορούμε να πούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν ε, υπογράφει ε, μια συμφωνία που δίνει προτεραιότητα ε, σε στόλο ενός κράτους μέλους δεν μπορεί να το κάνει εις βάρος του ελληνικού ευρωπαϊκού στόλου γιατί δεν ξέρουμε τι ιδιωτικές συμφωνίες έχει υπογράψει η Μαυρετανία. Επίσης, για τα κεφαλόποδα ιδιαίτερα ισχύουν αυτές οι ιδιωτικές συμφωνίες. Τώρα, για την βιωσιμότητα. Θα πρέπει να ενημερωθούμε για την πραγματική κατάσταση των αναλευτικών αποθεμάτων. Γιατί πρόκειται για μια συμφωνία που περιορίζει την πρόσβασή μας στους πόρου. Οπότε, ποια θα είναι η αντιπαροχή για τη μείωση αυτή. Θα πρέπει να μειωθεί αντίστοιχα και η αντιπαροχή. Αντίθετα, βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί η αντιπαροχή και έχουν αυξηθεί και οι διοικητικέ διατυπώσει Επίσης ε, ε, προστίθενται έλεγχοι ή προ... Ε, προστίθεται μια υποχρέωση για τον εφοδιασμό με καύσιμα και άλλα τεχνικά μέτρα που δεν συμβάλλουν στη βιωσιμότητα, απλώς ενισχύουν και επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο ενισχύουν το άχθος και επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις που θα πρέπει να καταβάλουν ακόμη μεγαλύτερες οικονομικές προσπάθειες. Δεν είναι λοιπόν ικανοποιητική η ελευτική συμφωνία. Θα πρέπει να εξετάσουμε τι τεχνικέ προποθέσει και αυτέ να ισχύουν για όλου του αλληλεί, οποιοδήποτε αλληλευτικού στόλου, εφόσον ε, στη συγκεκριμένη περιοχή. Θα πρέπει να είναι ισότιμοι λοιπόν όλοι οι αλληλεί. Και επίση να λάβουμε υπόψη την τομεακή ανάπτυξη. Γιατί η τομεακή ανάπτυξη αλληλεύει μειώνεται με βάση τη συμφωνία αυτή ούτε μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι οι μαυριτανικές αρχές δεν θα εκμεταλλευτούν την κατάσταση και τη, τα κονδύλια για την ανάπτυξη της αλίας. Τώρα, το θέμα των κεφαλόποδων είναι αυτό που επηρεάζει περισσότερο την δική μου περιφέρεια, τη Γαλλικία. Σε προηγούμενη συνεδρίαση είχαμε εγκρίνει την έκθεση για τη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής της κυρίας Ρόντουστ. Εκεί είχε πει ότι η αρχή της προφύλαξης θα πρέπει να έχει κάποια όρια. Και αν ακολουθούσαμε τους κανόνες της κυρίας Ρόντους, σε καμία περίπτωση δεν θα ε, καταλήγαμε σε συμφωνία που ουσιαστικά παροπλίζει 24 ελευτικά σκάφη. Γιατί εκεί υπήρχε ένα όριο με βάση την αρχή της προφύλαξης, της πρόληψης. Δεν μπορούμε να περάσουμε από το όλο στο τίποτα, από τον ένα χρόνο στον άλλον. Επίσης, τι, γίνεται, τι ξέρουμε από την κατάσταση του παρελθόντος. Έχουμε την, την μελέτη του 2013 που παραπέμπει στο 2012. Επίσης ε, γίνεται η παραπομπή στην συνεδρία του Αγαδίρ του 2010. Τα τελευταία στοιχεία που έχουμε μιλάνε για το 2009. Εκεί αναγνωρίζεται η διανοδική τάση των ε, αποθεμάτων. Βέβαια, διαπιστώνουμε υπάρχει ένας αλληλευτικός στόλος μικρής κλίμακας και φυσικά στηρίζουμε την ανάπτυξη ε, την ανάπτυξή του, αλλά έχουμε 200 μηχανότρατες ψυγεία με σημαία Μαυριτανίας που ουσιαστικά είναι ε, ιδιο, ιδιοκτησίες άλλων χωρών. Χρησιμοποιείται λοιπόν αυτός ο μηχανισμός όχι για να προστατευτεί ο, τοπικ, ντόπιο στόλος, αλλά για να διεισδύσουν άλλοι στόλοι στην εκμετάλλευση των πόρων. Και μάλιστα το Μάιο του 2011 είχαμε ένα ψήφισμα για το θέμα αυτό και μάλιστα στις 6 Ιουνίου, εκεί που διαπιστώναμε εμείς υπερεκμετάλλευση, με βάση στοιχεία του παρελθόντος, λέμε ότι θα πρέπει να μειωθεί, όχι να ε, καταργηθεί πλήρως η δραστηριότητα του κλάδου στην περιοχή. 6 λοιπόν Ιουνίου η Μαυριτανία συνάπτει συμφωνία με Κινέζικη εταιρεία για τα κεφαλόποδα. Αυτό μας φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση και μάλιστα ούτε συμβάλλει με τη δική μας ε, θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε με την κατάσταση των ε, αλληλευτικών αποθεμάτων. Γιατί αποκλείται μεν ο αλληλευτικός στόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα κεφαλόποδα, αλλά ταυτόχρονα δίνονται αλληλευτικές άδειες στα σκάφη μιας ιδιωτικής ε, κινέζικης εταιρείας. Μάλιστα πριν από λίγε μέρες ε, φαίνεται ότι αναστάλησαν αυτέ οι άδειε. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται στι επικρίσει που άσκησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη στάση τη μαυριτανικής κυβέρνηση. Αλλά μα ενδιαφέρει να έχουμε τα στοιχεία για αυτέ τι ιδιωτικέ συμφωνίε. Εμεί θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει σωστή αξιολόγηση του αποθέματος, να γίνει άμεση αξιολόγηση των αποθεμάτων, γιατί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σε μια κατάσταση όπου 20-30 ευρωπαϊκά σκάφη που ασχολούνται με τη δραστηριότητα αυτή έχουν καταδικαστεί ε, σε ανεργία και μάλιστα εξοβελίστηκαν από την περιοχή χωρίς καν σταδιακή μείωση ούτε καν πρόσφατη αξιολόγηση των αλληλευτικών αποθεμάτων, κάτι που είναι απαράδεκτο και ζητούμε άμεση αναθεώρηση αυτής της κατάστασης ήδη μεταβατική εφαρμογή της, το ανώτατο του ορίου για την αρχή της προφύλαξης και φυσικά γενική αναθεώρηση της συμφωνίας. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να την υποστηρίξουμε. Αλλιώ έχουμε πολύ σοβαρούς ενδιασμούς και επιφυλάξεις και δεν θα μπορέσουμε να την εγκρίνουμε. Μας τελειώνει ο χρόνος, οπότε είστε συντομότατοι. Ο κύριος Ρωμέβα είναι ο ε, Ευχαριστώ. Θα είμαι και εγώ λακωνικός. Εμένα με ενδιαφέρει κυρίω η απάντηση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα επίσης να επαναλάβω αυτά που είπε πριν ο Κρήτονας Αρσένης και συμφωνώ μαζί του. Έχουμε μια συμφωνία, η πρώτη φορά μάλιστα που έχουμε μια συμφωνία, όπου τηρούνται πολλές από τις αρχές που θέσαμε στο ψήφισμα και ίσως δημιουργηθεί ένα καλό προηγούμενο για σωστή συζήτηση και για τις επόμενες συμφωνίες. Θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό, ότι για πρώτη φορά γίνονται τα πράγματα όπως το ζητήσαμε εμείς, από πολλές απόψεις. Τρίτον, πάλι πολύ σύντομα θα ήθελα να πω ότι αντιλαμβάνομαι το θέμα του χταποδιού είναι πολύ ευαίσθητο και αφορά πολλά σκάφη και πολλούς αλληλευτικούς στόλους. Ακούσαμε τους εκπροσώπους των αλλιέων της Μαυριτανίας και νομίζω ήταν πολύ καθαρή και εξάστερη. Μα είπαν το θέμα του χταποδιού θέλουν να αποκλειστεί από τη συμφωνία, οπότε εμεί δεν έχουμε να πούμε πια τίποτα για αυτό το θέμα. Αυτή είναι η κυριαρχική βουλή τη Μαυριτανία. Δεν υπάρχει καν περιθώριο για συζήτηση. Και έχω την εντύπωση και διορθώστε με αν κάνω λάθο μετά την ακρόση που είχαμε με τους εμπειρογνώμονες, έχω την εντύπωση ότι δεν έχουμε ε, μεγάλο περιθώριο λιγμών για ένα εναλλακτικό σχέδιο, γιατί μερικοί ζήτησαν αναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Μαυριτανίας. Αλλά εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα για αναδιαπραγμάτευση. Δεν υπάρχει καν ένα διαπραγματευτικό περιθώριο. Θα ήθελα να μου το επιβεβαιώσει αυτό, παρακαλώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Λεβίν. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. θα ήθελα να απηχήσω τα μόλις υποθέντα ότι οι Μαυριτανοί υπήρξαν σαφέστατοι. Η κατηγορία των κεφαλοπόδων, του χταποδιού, είναι το μέσο να χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι. Και το ότι κατάφεραν να κάνουν να την κυβέρνηση να τους ακούσει είναι κάτι που πρέπει να υποστηρίξουμε. Και προχώρησαν και άλλο ένα βήμα αφαίρεσαν τις άδειε από τις κινέζικες στράτες. Αυτό είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα. Και νομίζω ότι και το Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίξαμε αυτό το σημαντικό βήμα για τους Μαυριτανούς αλληλείς. Ακριβώς αυτό θέλαμε να πετύχουμε όσον αφορά την εξωτερική διάσταση της αλληλευτικής μας ε, πολιτικής. Όπως είπε και ο κ. Ρωμέβα, είναι λάθος να πιστεύουμε ότι είναι δυνατή μια αναδιαπραγμάτευση. Σε όλα τα περιοδικά του κλάδου βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφοροι εμπλεκόμενοι φορείς που επιθυμούν πρόσβαση στα δυτικοαφρικανικά ύδατα, γυαλία. Και πριν μερικές εβδομάδες είδα ένα άρθρο για τη νέα ρωσική πολιτική. Οι Ρώσοι πραγματικά ψάχνουν να βρουν αλλιευτικές ε, δυνατότητες στη Δυτική Αφρική. Αν δεν κυρώσουμε αυτή τη συμφωνία, πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα άνοιγε την πόρτα για άλλους λιγότερο υπεύθυνου εμπορευόμενους που δεν έχουν ε, την αρχή της βιωσιμότητας που στηρίξαμε στο Κοινοβούλιο. Και υποστηρίζει και το Συμβούλιο. Το είδαμε στη συμπεράσματα του Συμβουλίου όσον αφορά την εξωτερική πολιτική. Το Συμβούλιο είπε ναι στη συμφωνία και στην κύρωση αυτής και θα πρέπει να κάνει το ίδιο το Κοινοβούλιο, κατά την άποψή μου. Και κάτι άλλο πολύ καλό που έχει για αυτή η συμφωνία είναι η ρήτρα περί μη διάκρισης που δεν ανέφερε ο κύριος Μάτο. Λέει ότι όλες οι τρίτες χώρες που θέλουν να αλλιεύουν στα μαυριτανικά ύδατα θα πρέπει να εφαρμόζουν τους ίδιους τεχνικούς κανόνες και περιορισμούς όπως και ο στόλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και έτσι όλοι οι άλλοι στόλοι ε, σπρώχθηκαν στα πιο ανοιχτά από τις παράκτιες περιοχές. Πήγανε στα 20 ναυτικά μίλια. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό διαπίστωσα όταν διάβαζα τις ειδήσεις προάλλες για τον πόλεμο στο Μαλί. Ε, ξέρουμε ότι είναι παρούσα στην περιοχή και η Αλκάιντα. Είναι πολύ ευαίσθητη η χρονική στιγμή, ευαίσθητη ιστορικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα κάνει καλό στα συμφέροντά της αν ε, ταράξει τους ντόπιου πληθυσμού της περιοχής τώρα. Ούτε τώρα ούτε ποτέ, αλλά ειδικά τώρα ε, πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να φαίνεται ότι είναι υπεύθυνος εταίρος ε, είναι εταίρος με την πραγματική έννοια του όρου και ελκυστικός εταίρος στο μέλλον όσον αφορά την αλληλεία και για άλλους τομείς. Αυτό είναι και το πλεονέκτημα που θα μπορούσε να έχει, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι Ρώσων, Κινέζων, Κορεατών που δεν τους εκτιμούν τόσο. Όπως μας είπε και ο πρόεδρος Αχμέτ, εκπρόσωπος του ευτικού τομέα, λέει ότι είναι ευπρόσδεκτη η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ότι ήμασταν πολύ σωστοί στις διαπραγματεύσεις και αυτό θα πρέπει να το εκτιμήσουμε. Και αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρνηθεί την κύρωση της συμφωνίας, αυτό θα ήταν τεράστιο σφάλμα όσον αφορά την εικόνα μάλιστα της Ευρωπαϊκής Ενώσης στην περιοχή. Ευχαριστώ. Η κυρία Μιράντα, επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ. Μία τέτοια συμφωνία θα πρέπει να είναι δίκαιη για όλους. Το επαναλάβαμε. Δίκαιη, χωρίς ε, διακρίσεις. Ίση για όλους. Δίκαιη για όλα τα συμβαλώμενα μέρη, όχι μόνο για το ένα συμβαλόμενο μέρος. Και αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο που δεν έχει τηρηθεί. Το πρωτόκολλο δεν εξασφάλισε ούτε συμμετοχή του κλάδου, ούτε έλαβε υπόψη την κοινωνική διάσταση, ούτε έλαβε υπόψη τις κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες ε, του αποκλεισμού ενός τμήματος του ελευτικού στόλου. Θα είναι τεράστιος ο αντίκτυπος στην απασχόληση, όχι μόνο για τον ελληνικό στόλο των κεφαλόποδων της δικής μου πατρίδας, αλλά θα έχει επιδράσεις και στο στόλο της Μαυριτανίας, σε ό,τι αφορά τα πληρώματα των μαυριτανικών σκαφών. Ή μήπως θα έχουν καλύτερες ε, εργασιακές συνθήκες, κοινωνικές και οικονομικές με το κινέζικο στόλο από ό,τι με το δικό μας. Δεν νομίζω. Τέλος. Για τη ζώνη αποκλεισμού και τα μίλια. θεωρώ ότι ο στόλος των κεφαλόποδων και η παράκτη αλία ε, δεν ε, είναι αντιφατικές μεταξύ τους. Πιστεύω ότι μία αλληλευτική συμφωνία και ένα πρωτόκολλο θα πρέπει να είναι δίκαιο για όλους, το επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά. Θα πρέπει να είναι δίκαιο και για τους ε, παράκτιους αλληλείς ε, μικρής κλίμακας της Μαυριτανίας, αλλά και για μας. Επαναλαμβάνω, η παράκτη αλληλεία μικρής κλίμακας της Μαυριτανίας θα πρέπει να υποφελείται από καλές συνθήκες, από καλές εγκαταστάσεις, από τρόπο που θα τους ευνοεί ε, η συμφωνία, αλλά θα πρέπει αντίστοιχα πρόσφορες να είναι οι συνθήκες και για, του, για τους Ευρωπαίους αλείς. Όχι να τους τριμώχνουμε ε, και να τους επιβάλλουμε άνισα και δυσβάσταχτα μέτρα. Εκπροσωπώ τους συμπατριώτες μου και νομίζω ότι αυτό το συμφέρον θα πρέπει να προτάξω εδώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε και μια ευαισθησία για θέματα ανάπτυξης μια ευαισθησία για τους λιγότερο ευνοημένους ε, λαούς άλλων χωρών. Αλλά θα πρέπει να είμαστε δίκαιοι σε κάθε περίπτωση. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κοινωνικό αντίκτυπο πολύ αρνητικό. Γύρω στις 500 μόνο στην ζώνη του Αμοράσου. Δεν έχουμε ελευτικές ζώνες, τα σκάφη μένουν αγκυροβολημένα, δεν έχουν εναλλακτικέ ε, λύσεις. Πάνω από 400 ναυτικοί βρίσκονται στην ξηρά, και επαναλαμβάνω, η ζώνη της Ευρώπης από την οποία κατάγομαι εξαρτάται αποκλειστικά από την αλία. Γι' αυτό υφίσταται πολύ δυσμενή συνέπειες από τη συμφωνία αυτή. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλην πληρώσει το αντιστάθμισμα με χρήματα των φορολογουμένων να ζητήσει κατ' επίγουσα σύγκληση της ΕΤΟΕΑ και της Μικτής Επιτροπής να αξιολογήσει την κατάσταση των αποθεμάτων και κυρίως ε, να αντιμετωπίσει δίκαια και ισότιμα ε, κάποιους πληθυσμούς που εξαρτώνται από την αλία πλήρως όπως είναι η Γαλλικία. Στην Επιτροπή όλοι θέλουμε συμφωνία, αλλά κυρίως δίκαιη για όλους και μια συμφωνία με τους όρους ε, που έχει αυτή τη στιγμή θα πρέπει να απορριφθεί. Γιατί δίνει λιγότερες αλληλευτικές δυνατότητες πληρώνοντας περισσότερα χρήματα. Επαναλαμβάνω, η Μαυριτανία έχει δικαίωμα να χαράξει τη δική της αλληλευτική πολιτική. Αν ε, συνάψει όμως μια αλληλευτική συμφωνία και θέλει σύμπραξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα πρέπει να γίνει αυτό στην πλάτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην πλάτη των φορολογουμένων, στην πλάτη των άνεργων ψαράδων, γιατί εκατοντάδες ε, ψαράδες ε, και άλλοι εργαζόμενοι θα μείνουν άνεργοι σε ζώνες που εξαρτώνται αποκλειστικά και μόνο από την αλία και δεν έχουν ε, άλλη λύση. Και θα ήθελα να καλωσορίσω εκπροσώπους από τη Γαλλικία που ασχολούνται με την αλία κεφαλοπόδων. Έξι μήνες τώρα ζουν με επιδόματα και ήρθαν εδώ για να ακούσουν τη συζήτηση και να ακούσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί δεν άκουσε και τη δική τους φωνή, γιατί δεν τους εμπεριέλαβε στις διαβουλεύσεις. Επαναλαμβάνω, μια συμφωνία με αυτού του όρου θα πρέπει να απορριφθεί. Λέμε όχι, θέλουμε δίκαιε συμφωνίε για όλου. Ευχαριστώ. Ε, η κυρία Φράγκα είναι η επόμενη απολύτρια. Sí. Bueno, yo, como Ευχαριστώ. Αυτή τη φορά θα είμαι πιο σύντομη, μια και τα είπα και προηγουμένω. Νομίζω θα πρέπει να υπάρχει μια βρότητα στι επιχειρηματολογίε, ιδιαίτερα για το οχταπόδι στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό που λέγαμε για το χταπόδι είναι ότι υπάρχει υπερεκμετάλλευση και γι' αυτό θα πρέπει να εφαρμοστούν διαφορετικές διατάξεις στο πρωτόκολλο για το χταπόδι ειδικά. Τώρα, τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν ε, για το ψήφισμα αυτό ήταν στοιχεία του 2008, ενώ τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν βελτίωση της κατάστασης του αποθέματος. Τώρα αλλάζουμε την επιχειρηματολογία και λέμε τώρα το πρόβλημα δεν είναι η υπερεκμετάλλευση, είναι θα πρέπει να αφήσουμε την απόλυτη εκμετάλλευση του ελευτικού πόρου του χταποδίου στη Μαυριτανία. Ναι, η Μαυριτανία να κάνει τι θέλει με τα αλληλευτικά της αποθέματα. Το θέμα το όμως είναι ότι στο αλληλευτικό πρωτόκολλο υπάρχει μηδενικό τάκ, για τα κεφαλόποδα που εξαρτάται από τη βελτίωση του αποθέματος και όχι από την αποκλειστική εκμετάλλευση από τη Μαυριτανία. Υπάρχει μία ειδική κατηγορία μηδενικό τάκ για τα κεφαλόποδα στον αλευτικό πόρο. Προσοχή λοιπόν να ξέρουμε με σαφήνεια τι έκανε και για ποιο λόγο το έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και από τη στιγμή που υπάρχει μηδενικό τάκ για τα κεφαλόποδα που εξαρτάται από την κατάσταση των πόρων, από τη στιγμή που βελτιωθεί το ελευτικό απόθεμα, τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα προβλέψει ΤΑΚ και σε ό,τι αφορά τη, νέα διαπραγμάτευση ή την αναδιαπραγμάτευση. Ε, όπως είπε ο κ. Δεπιπέρ, ε, είναι έτοιμοι να κάνουν κάποιες ε, βελτιώσεις ε, στη μεικτή Επιτροπή. Ε, ταυτόχρονα ο κύριος Ντεμπιπέρ είπε ότι αυτή η συμφωνία ήταν η καλύτερη δυνατή και ότι δεν επιδέχεται αναδιαπραγμάτευση. Δεν ξέρω. Άλλα λέει ε, ιδιωτικά και άλλα λέει δημόσιο ο κ. Ντεμπιπέρ. Τι θα κάνει τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα κάνει τίποτα στη μεικτή επιτροπή, γιατί ακούγονται αντιφατικά σχόλια. Από τη μια λέει θα βελτιωθούν οι τεχνικέ προποθέσει στη μεικτή επιτροπή και από την άλλη λέει ότι είναι η καλύτερη δυνατή συμφωνία και δεν επιδέχεται αναδιαπραγμάτευση. Τέλο, να πω ότι μια συμφωνία 70 εκατομμυρίων όταν αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο 7 σκάφη που αλλιεύουν στην περιοχή, τι να σας πω, όπως είπε και ο προλαλής σας, δεν είναι εμπορική αυτή η συμφωνία. Μόνο όταν 3 εκατομμύρια είναι αναπτυξιακή βοήθεια, να, ε, να πληρώνουμε 70 εκατομμύρια όταν μόνο 7 σκάφη αλλιεύουν είναι υπερβολικό. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Μπιλμπάου, επόμενη. Ευχαριστώ. Πριν ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα να θέσω και εγώ δύο ερωτήσει. Αφού ακούσαμε τον κλάδο και τους εκπροσώπους ε, των, των διαφόρων πολιτικών ομάδων, θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρεί ε, σκόπιμο να κάνει μια διεξοδική ανάλυση της κατάστασης του αποθέματο του χταποδιού. Ή, ε, και δεύτερο, θεωρεί ότι ε, θα πρέπει να επιληφθεί και πάλι η μεικτή επιστημονική επιτροπή. Γιατί αν δεν συγκληθεί η Μικτή Επιτροπή και αν δεν είναι διατεθειμένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αναδιαπραγμάτευση, θα ήθελα να μας πει, έχει σταθμίσει τις αρνητικέ συνέπειες που θα έχει για τον κλάδο η εφαρμογή αυτού του πρωτοκόλου. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη 1.200 άνεργους λόγω της αλληλευτικής συμφωνίας. Και αναμένονται νέες απολύσεις, και άλλες επιχειρήσεις που θα κλείσουν, Οπότε, έχοντας όλα αυτά τα στοιχεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποια στρατηγική θα εφαρμόσει και τι διέξοδο ε, θα προτείνει για τα ληφτικά αυτά σκάφη που δεν μπορούν να ψαρεύουν πια πουθενά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έβαλα και εγώ το όνομά μου στον κατάλογο. Ξεκινώ με μια ομολογία την παρέμβασή μου. Συνήθως στις εξομολογήσεις Λες είμαι ένας φτωχός και αμαρτωλός άνθρωπος. Η τελευταία συνεδρία της Επιτροπής Αλληλείας διέπραξε τα κάτω θυσφάλματα. Είχα ένα μικρό κόκκινο αριθμό, ένα, ένα ε, Είπα, μου έλεγε ο διάβολος αριστερά μου, ε, ας πάμε για τη συμφωνία, θα ψαλεύουμε μερικά ε, χρόνια και θα επιστρέψουμε στι διαπραγματεύσει με προσαρμοσμένη άποψη. Προσπάθησα όμως να είμαι καλός και αγαθός. Άρα πρέπει να υπερψηφίσουμε τη συμφωνία γιατί όλες οι άλλες επιλογές είναι αρνητικές. Αν εξετάσει κανείς τα επιχειρήματα, βλέπει ότι υπάρχουν πολλά επιχειρήματα υπέρ της συμφωνίας. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν θέλουμε να πούμε τι θα έπρεπε να κάνει η Μαυριτανία. Είναι ολιστηρός ο δρόμος να το εξετάσει κανείς το θέμα από ηθική σκοπιά. Υπάρχουν πολλά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα στην Ευρώπη και πρέπει να τα φροντίσουμε. Γύρω από αυτό που περιεστράφει η συζήτηση αλλά να λύσουν τα προβλήματα μέσω της Ελληνική συμφωνίας με τη Μαυριτανία. Λάθος είναι αυτό. Οπότε θα είμαι λακωνικός αν υποσχεθεί και ο Κρίς να είναι έτσι συντομότερος. Ευχαριστώ. Πράγματι, Πρόεδρε, και ζητώ συγγνώμη περίμενα, στο, περίμενα πολλή ώρα στο διάδρομο απογείωσης. Έτσι είναι η ζωή στη Βρετανία, ο Πρόεδρος. Δεν είμαστε τόσο καλά οργανωμένοι όπως οι Φιλανδοί, λέει ο μιλητής. Εκφράστηκαν ανησυχίες. Δεν πετυχαίνουμε πολλά για τα χρήματα που δίνουμε. Ίσως αναφέρθηκε αυτό. Ποιο είναι το περιβάλλον του ανταγωνισμού. Να μας πει η Ευρωπαϊκή Επίτροπη, αν δεν είμαστε εμείς, ποιος θα συνάφει τη συμφωνία, ποιος θα πληρώσει για την αλία. Ξέραμε ποιοι άλλοι ενδιαφέρονται. Μας ξεγέλασαν, μας την παίξανε, είμαστε, είναι καλή συμφωνία για μας. Αυτό θέλω να ξέρω. Ευχαριστώ λέει πρόεδρος και κλείνει το μικρόφωνο του. There are Πολλές ερωτήσεις για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κ. Μπέρκ μπορεί να απαντήσει. και από εκεί πέρα βλέπουμε τι θα κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόκληση να απαντά κανείς σε ένα σύνολο ερωτήσω. Να μην μπω στην επίθεση που δεχτήκαμε όσον αφορά το πρωτόκολλο αυτό, την συμφωνία με τη Μαυριτανία. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Όλοι έχουμε επίγνωση της σημασία των διακυβευμένων που συζητούνται σήμερα εδώ. Διακυβεύματα λοιπόν που αφορούν τον Ευρωπαϊκό Στόλο αφορούν τη Μαυριτανία και τα κράτη-μέλη. Δεν αφορά μόνο ένα ή δύο κράτη-μέλη που αλλιεύουν στη Μαυριτανία, δωδεκα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να ψαρέψουν. Υπάρχει και γενική πτυχή, ξέρουμε όλοι τι αντίκτυπο μπορεί να έχουμε για κάποιες περιοχές όπως είναι τα Κανάρια νησιά και η Γαλλικία. Το πρωτόκολλο που διαπραγματευτήκαμε και μονογραφήσαμε σίγουρα είναι ατέλες. Συμφωνεί όμως με την δοθήσα διαπραγματευτική εντολή που μας το Συμβούλιο. Και συνάδει και με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίως όσον αφορά τα κάτωθη. Τον περιορισμό της αλευτικής δραστηριότητα το πλεόνασμα το αλευτικό και λαμβάνεται υπόψη το αλευτικό απόθεμα. Κάποια αποθέματα που ήταν στο προηγούμενο πρωτόκολλο ήταν αντικείμενο υπερεκμετάλλευσης ή τα είχαμε εκμεταλλευτεί πλήρω. Έγινε αυτή η τα ειχαμε εκμεταλλευτει πλήρω. εγινε αυτη η αποτιμηση το θύμισαν οι πυρογνώμονε. Είναι μια διαπίστωση την οποία κάναμε ότι δεν ήταν βιώσιμο το προηγούμενο πρωτόκολλο και χρειαζόταν ιδέουσα προσαρμογή. Λάβαμε υπόψη διαπραγματεύσει και τετήματα των Μαυριτανών όσον αφορά τον στόλο αλίας μικρής κλίμακας και ο πρόεδρος ζήτησε να έρθει ο πρόεδρος εδώ των αλιέων για να αναφερθεί και να δει πόσο σημαντική είναι να απελευθερωθεί αυτή η αλληλεία για τους ντόπιου αλίες. Η συνέπεια σε τοπικό επίπεδο έπρεπε να ληφθεί υπόψη. Και ήταν στο επίκεντρο των ε, όσων ζητούσαν οι Μαυριτανοί. Έχουμε συντονιστεί, εφαρμόσαμε την αρχή της μεταρρύθμισης, κάτι που δεν αναφέρθηκε σήμερα. Αυτή η ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πάντα παρούσα σε όλες τις ελευτικές συμφωνίες και συμπεριλαμβάνεται και στο πρωτόκολλο που συζητούμε τη Μαυριτανία. Και τέλος υπάρχει ένα άρθρο σημαντικό κατά την άποψή μας. Το πρώτο, σημείο 4, που επιμένει επί της προτεραιότητας πρόσβασης των ευρωπαϊκών στόλων και αυτό είναι σημαντικότατο. Και Φανίζεται και σε διάφορους τομείς αλληλευτικούς όπως τα πελαγικά είδη. Θα επανέλθω αργότερα σε αυτό, με διευκρινήσεις για τους διάφορους τομείς που καλύπτει η συμφωνία. Πριν το κάνω αυτό, να αναφερθώ σε κάτι που εθίγει επανειλημμένα. Το κόστος της συμφωνίας και το επίπεδο της οικονομικής αντιστάθμισης όσον αφορά τη συμφωνία αναφέρθηκε ότι είναι πολύ ακριβή συμφωνία σε σχέση με τις δυνατότητες αλληλευτικές που δίδονται στους Ευρωπαίους. Να υπενθυμίσω εδώ κάποια πράγματα, πραγματικά στοιχεία, προφανή. 76 εκατομμύρια με 70% πήγαμε ε, όσον αφορά την συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δεν, είναι, δεν έχει μειωθεί όμως η ελευτική προσπάθεια συνολικά. Έχουμε τάκ 0 για τα κεφαλόποδα βέβαια, αλλά μίλης μονούμε ότι για τα πελαγικά είδη από 250.000 τόνους πάμε στους 300.000 τόνους. Διατίθενται αυτά τα είδη ε, μεγαλύτερες ποσότητες για τα πελαγικά είδη από ό,τι κατά την παρελθούσα συμφωνία. Από τα 250.000 στα 300.000 περάσαμε. Υπάρχει περαιτέρω δυνατότητα, αλλά πρέπει να καταβληθεί και ένα τίμημα. Όταν συγκρίνουμε τις δυνατότητες που υπήρχαν και θα υπάρξουν πρέπει να λάβουμε υπόψη έχω τον παράγοντα. Να πω επίσης ότι όσον αφορά την περίοδο του περασμένου πρωτοκόλου, 2007 α πάρω σαν έτο αναφορά, αυξήθηκαν οι τιμέ. Αν δούμε τα πελαγικά είδη, έχουμε αύξηση περίπου 15% κατά την περίοδο 2007-2011. Και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όσον αφορά την αποτίμηση αξία τη συμφωνία και όσον αφορά τη σύνθεση των αλλιευμάτων. Ο διαχωρισμό σε ζώνε των πελαγικών ειδών από τα 13 μέχρι τα 20 ναυτικά μίλια, αυτή η απόσταση έχει σαν συνέπειε να στοχεύονται περισσότερα τα είδη που έχουν μεγαλύτερη αξία. Όπω είναι ο Βαγκαλιάρο σε σχέση με τη σαρδέλα και την φρίσα. Αν πάρουμε τη μέση τιμή για τα πελαγικά είδη 600 ευρώ τον τόνο, κάτι που αναφέρθηκε προηγουμένω από αμπειρογνώμονα, αυτή η τιμή αφορά κυρίως τις αρδέλες και ε, την φρύσα. Στον τομέα για τα άλλα είδη, τα πιο ακριβά είδη, έχουμε, όπως τα σαυρίδια, έχουμε ψηλότερες τιμής. 200.000 ε, ε, ευρώ τον τόνο. Στις τιμές που πληρώνουμε υπάρχουν δύο συνισταμένε. Η μία είναι η εισφορά που πληρώνουν οι πλειοκτήτε, οι συναυλωτές. Η αύξηση είναι σημαντική, πιο μεγάλη για κάποια τμήματα του στόλου, όπω είναι για τα πελαγικά είδη. Προσπαθήσαμε συζήτηση, συζητήσει, διαπραγματεύσει να διαμορφώσουμε το επίπεδο των αυξήσεων, συναρτήσει των κατηγοριών των σκαφών και των διαφόρων χαρακτηριστικών ε, του κάθε στόλου. Η αύξηση ήταν υψηλή για τα πελαγικά, μεγάλη, λιγότερο μεγάλη για τα άλλα είδη σκαφών ε, που αλλιεύουν. Στις συζητήσεις τις πολλές που είχαμε με τον τομέα των πελαγικών ειδών δεν ήταν πρώτο μέλημα η τιμή. Ίσως το θέμα της απόστασης ήταν κάτι σημαντικό, τεχνικές λεπτομέρειες. Αλλά δεν ήταν η εισφορά που τους απασχολούσε ε, παραπάνω το πρώτο πρόβλημα όσον αφορά τη συμφωνία. Και τα στοιχεία που παρετέθησαν από τον κύριο Καγιάρ είναι ενδιαφέροντα πολύ διότι δείχνουν τα διάφορες φορές σε ποσοστά της αξίας των αλλιευμάτων. Θα σημειώσω το και εγώ για τη γαρίδα περίπου 8% εισφορά της αξίας του αλλιεύματος, για, τους, για τον τόνο 20% περίπου και εισφορά για τα πελαγικά είδη που είναι περίπου το 20% της αξίας του αλλιεύματος. Αυτά όσον αφορά την τιμή ε, της φρύσας χωρίς να λαμβάνουν υπόψη και τα τις περισσότερες τιμές, τις τιμές για τα σαφρίδια. Αυτά είναι κάποια στοιχεία οικονομικής φύσεως που ελπίζω αυτά τα στοιχεία δίνουν μια νέα ισορροπία στη συζήτηση. Αν επιτρέπετε να παραθέσω κάποια στοιχεία όσον αφορά τις διάφορες κατηγορίες των ηχθείων που αναφέρθηκαν στη συζήτηση. Θα ξεκινήσω από το πελαγικά είδη και μετά θα, θα αναφερθώ στις γαρίδες και μετά στα κεφαλόποδα. Όσον αφορά τα πελαγικά είδη είναι σαφές ότι υπάρχει ένα πρόβλημα υπερεκμετάλλευσης όσον αφορά την φρύσα. Οι μελέτες δεν ήταν σαφέστατες. Εμείς θέλαμε να εφαρμόσουμε την αρχή της πρόληψης και να μειώσουμε την αληφτική προσπάθεια όσον αφορά την φρύσα. Σημαντικό στοιχείο που υπενθυμίστηκε και από τον εκπρόσωπο τη Ομοσπονδία των Αλλιών τη Μαυριτανία είναι και του ενδιαφέρεται και ο τοπικό στόλο για την Φρύσα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη λοιπόν και αυτό το συναγωνισμό με ε, του εθνικού αλλιεί. Ε, Στι διαπραγματεύσει ε, σκεφτήκαμε να υπάρχει υποποσόστοση για την Φρύσα, αλλά το αρνήθηκε ο στόλο αυτό. Έπρεπε να καταλήξουμε σε μια, να αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη κατάσταση, έπρεπε να αλλάξει η στρατηγική για το στόλο από 13.000 να πάμε στα 20, στα 10, από τα 13 μίλια στα 20 μίλια από από τις Υπάρχουν στόλοι που μπορούν να ενταχθούν στα νέα δεδομένα. Υπάρχουν δύο βαλτικά σκάφη που αλλιεύουν τώρα στη Μαυριτανία. Άλλα τμήματα του πελαγικού στόλου δεν ακολούθησαν την ίδια στρατηγική, αλλά είναι σε θέση να προσαρμοστούν διόντως, ούτω ώστε να εκμεταλλευτούν τι 300.000 τόνου που είναι διαθέσιμοι. 300.000 τόνοι αντιστοιχούν ακριβώς στην ποσότητα που μας ζητήθηκε από τον τομέα. Και κάτι σημαντικό που αναφέρθηκε από κάποιους βουλευτές είναι οι τεχνικές ε, συνθήκες που εφαρμόζονται για όλους τους τόλους για τα πελαγικά είδη. Για τους Ρώσους, για τους Ουκρανούς, για τους Ασιάτες, ακριβώς οι ίδιες προδιαγραφές ισχύουν. Οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως και για τους ευρωπαϊκούς τόλους. Μετά υπάρχει μια σειρά κρίσεων που ακούσαμε όσον αφορά τεχνικές διατάξεις, δεν επισέθω πολλές λεπτομέρειες. Το θέμα της μεταφόρτωσης και εκφόρτωσης. Αυτές οι διατάξεις του πρωτοκόλου περιορίζονται από, τις, από την επιμελητία και από το κόστος, από τους υλικούς περιορισμούς. Κάποιες μεταφορτώσεις θα λάβουν χώρα, αλλά πιθανότατα στο μέλλον οι εκφορτώσεις θα λαμβάνουν χώρα στον Αντιμπού για να απευθυνθούν μετά προς την Λασπάλμας. Ε, όλες οι ενδείξεις που έχουμε, όλες τις επαφές που είχαμε τους Μαυριτανούς μας δείχνουν ότι δεν υπάρχει μεταπητική βιομηχανία και επαρκή αγορά στη Μαυριτανία για να επεξεργαστεί τέτοιε ποσότητε ε, ψαριών. Εγώ δεν θα ανησυχούσα πολύ για το πόσο θα επηρεάσει αυτή η δραστηριότητα τη Λασπάλμα το θέμα του μονοπωλίου για τον ε, εφοδιασμό σε καύσιμα είναι κάτι που αναφέρθηκε στο, στην παρουσίαση του κ. παρόλο που δεν περιλαμβάνεται στο πρωτόκολλο. Μάθαμε ότι αυτό το μονοπόλιο καταργήθηκε. Αυτό είναι καλό για το στόλο. Αναφέρθηκαν και κάποιες υποχρεώσεις, κάποιες δωρές, ε, κάποιες χρηματοδοτήσεις. Αυτά ήδη προβλεπόταν και στο προηγούμενο πρωτόκολλο ίσως δεν είχαν επισημοποιηθεί, αλλά ήταν κάποιες υποχρεώσεις, κάποιες αντισταθμίσεις ε, που έπρεπε να δώσει ο στόλος. Για τα πελαγικά είδη είμαστε πεπισμένοι ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη συμφωνία. Είναι θέμα αλλαγής στρατηγικής, ίσως και βούλησης και εν πάση περιπτώσει η άσκηση αλληλευτική δραστηριότητα είναι δυνατή υπό του όρου που προβλέπει το πρωτόκολλο, υπό τον όρο ότι αν υπάρξουν προφανεί δυσκολίε, Γι' αυτό πρέπει, για να το δει κανεί πρέπει να πάει να ψαρέψει. Θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Θα πρέπει να πάμε να συνομιλήσουμε με τους Μαυριτανούς συνομιλητές. Είναι πρόθεσή μας να διοργανωθεί μια μεικτή επιτροπή πολύ γρήγορα ε, με τη συμμετοχή των Μαυριτανών. Όσον αφορά τα οστρακοειδή και τις γαρίδες, και εκεί άλλαξε, άλλαξαν οι ζώνες, που έχει, κάτι που έχει συνέπειε για το στόλο, κάτι δικαιολογημένο λόγω τη αρνητική συνέπειας που έχει αλία, που θα μπορούσε να έχει αυτή η αλία, ε, υπό του όρου του προηγουμένου πρωτοκόλου. Καταφέραμε να πετύχουμε συμβιβασμό 50% των, των σκαφών μπορούν να πάνε, ψαρεύσουν μεταξύ 6 και 8 ναυτικών μιλίων. Είναι πιο δύσκολη η αλία, είναι πιο επαχθής ο κύκλος, αλλά είναι δυνατόν να γίνει αυτή η αλία υπό τους όρους του πρωτοκόλλου και σε επαφές που είχαμε με Βρετανούς είδαμε ότι υπάρχει από την πλευρά του άνοιγμα να συζητήσουν τις τεχνικές προϋποθέσεις ε, για αυτή την αλληλεία, το επίπεδο ε, των παραλιευμάτων που θα πρέπει να ε, επιβάλλεται στα λευτικά σκάφη που αλλιεύουν γαρίδε. Τόσο αφορά τα κεφαλόποδα, να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν βρετανικά σκάφη που αλλιεύουν τώρα τα κεφαλόποδα Ήδη αναφέρθηκε πιστεύω, δεν υπάρχουν σκάφη κινέζικα υπό άλλη σημεία. Αυτή η αλία αφορά μόνο στα σκάφη που έχουν μαυριτανική σημαία. Είναι απόφαση της κυβερνήσεως. Έκανε αυτή την επιλογή και δίνει αυτό το προνόμιο στους εθνικούς αλείς και θα πρέπει να το σεβαστούμε αυτό σαν μια απόφαση κυριάρχου κράτους. Πρέπει να ληφθεί υπόψη. Μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Υπάρχουν δύο πτυχές. Υπάρχουν τα αποθέματα από τη μια και οι πολιτικές αποφάσεις από την άλλη και το πλαίσιο των σχέσεων με κάποιες ε, κινέζικες εταιρείες. Πράγματι το απόθεμα των κεφαλοπόδων μπορεί να αλλάξει πολύ γρήγορα. Είναι ένα είδος που έχει ένα σύντομο κύκλο ζωής και αναπαραγωγής. Τα πράγματα σίγουρα θα βελτιωθούν, διότι σταματήσαμε την αλία των κεφαλοπόδων από τον Αύγουστο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι είμαστε διαθέσιμοι, μπορούμε να εξετάσουμε εκ νέου σε επαφέ βέβαια με του Μαυριτανού, ποια είναι η κατάσταση των αποθεμάτων με πρόσφατα στοιχεία, ούτω ώστε να επικαιροποιήσουμε τα επιστημονικά δεδομένα επί των οποίων βασιστήκαμε για τι διαπραγματεύσει του πρωτοκόλου. Η μελέτη του Ισπανικού Ινστιτούτου αναφέρθηκε επίση, τη Οκεανολογία. Το είπαμε επανειλημμένα. Είναι ένα μοντέλο διαχείριση που παρουσιάζει διάφορε υποθέσει ενδιαφέρουσε, που θα πρέπει όμω να επικυρώνεται και να διασταυρώνονται πληροφορίες με τους Μαυριτανούς. Εγώ μπορώ να σας πω ότι αφού επελήφθην του θέματος, έχουμε πρόθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διοργανώσουμε τάχιστη συνεδρίαση της ε, Μικτής Επιστημονικής Επιτροπής, τουλάχιστον από τώρα μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, ούτως ώστε πριν από τη συνεδρίαση της Μικτής Επιτροπής να γίνει η συζήτηση αυτή για να μπορούμε να έχουμε πρόσφατα στοιχεία στη διάθεσή μα, αξιόπιστα στοιχεία όσον αφορά τα αποθέματα των ε, κεφαλοπόδων. Και εν συνεχεία υπάρχουν και άλλε δύο πτυχέ. Η πολιτική, αν τα αποθέματα βελτιωθούν, η μαυριτανική κυβέρνηση θα δεχτεί να μα δώσει ένα ποσοστό του πλεονάσματο. Αυτή πρέπει να αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα απηχήσει, όπως συχνά το έκανε στις πραγματεύσει την άποψη αυτή για να δοθεί ένα ποσοστό των αποθεμάτων κεφαλοπόδων τουλάχιστον για να συντονιστούμε τι προτεραιότητε και τη κυβερνήσεως τη Μαυριτανίας και να συντονιστούμε και με τα συμφέροντα των τόπιων αλλιέων. Όσον αφορά το Μερλούκιο, ε, με ρωτήσατε γιατί βάλαμε στι 4.000 τόνου την ποσόστοση. Ε, τηρούμε το παλιό πρωτόκολλο, ήταν περίπου 3.600 τόνους. Προσπαθήσαμε λοιπόν να μην βλάψουμε κανένα και λάβαμε υπόψη την ε, χρήση του παρελθόντος, την πραγματική χρήση. Πριν είχαμε ποσόστοση που είχε διαφορετική προσέγγιση. Περάσαμε στο ΤΑΚ τώρα, από την προηγούμενη προσέγγιση, ε, και βασιστήκαμε στα ιστορικά στοιχεία. Τώρα, ποιος αλλιεύει στα ύδατα της Μαυριτανίας. 36 σκάφη αλλιεύουν που έχουν άδεια αλίευση ή είναι καθοδόν προς αδειοδότηση. Λίγο μεγαλύτερο αριθμός από αυτόν που αναφέρθηκε στη συζήτηση. Έχουμε δύο σκάφη για το μαύρο μπακαλιάρο και κάποια για τα βαθυπελαγικά. 20 περίπου σκάφη ε, για αλίευση τόνου. Και με παραγάδια και, ε, με, ε, και τράτες. Και δύο σκάφη πελαγικά της Λιθουανίας που έχουν ζητήσει άδεια και που δραστηριοποιούνται στα ύδατα της Μαυριτανίας. 36 σκάφη λοιπόν, από 122 συνολικά, περίπου το 1 τρίτο του στόλου που θα μπορούσε να λιεύσει ήδη βρίσκεται εκεί. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι το πρωτόκολλο συμφέρει κάποια κράτη-μέλη, κάποιους στόλους, άρνηση Κύρωση του πρωτοκόλλου θα έχει και αρνητικέ συνέπειε για αυτό το κομμάτι του ε, στόλου που ε, παρόλο που δεν ακούγεται τώρα εκμεταλλεύεται ήδη το πρωτόκολλο, πρωτόκολλο που εφαρμόζεται προσωρινά. Όλων αυτών λεχθέντων να σας ανακοινώσουμε ότι μια μεικτή επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει πιθανότατα στις 19 και 20 Φεβρουαρίου με τη συμμετοχή των Μαυριτανών. Εκεί με μεγαλύτερη λεπτομέρεια θα εξεταστούν κάποια σημεία και διάφορες τεχνικές ε, συνθήκες που συζητήθηκαν σήμερα και προϋποθέσεις χωρίς να λησμονούμε κανένα θέμα έστω και δύσκολο προτιθέμεθα αυτή η μεικτή επιτροπή να συνεδριάσει με τη συμμετοχή των Μαυριτανών να συζητήσουμε τη γενναλία της ε, γαρίδας των πελαγικών ειδών επίσης για τις διάφορες ζώνες και αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε και προτιθέμεθα να ε, μιλήσουμε και για τα παραλιεύματα, για το διαχωρισμό σε ζώνες, σε διάφορες κατηγορίες και για το καβούρι ε, και για τα καβούρια, κάποιες περισσότερες άδειε ίσως ή μεταφορά μεταξύ αδειών, ε, μεταξύ των ειδών σκαφών που αλλιεύουν τον τόνο, στρατών και σκαφών με παραγάδι, την χρήση και την απασχόληση των Μαυριτανών αλλιέων. Υπάρχουν διάφορα θέματα στην ημερήσια διάταξη και το θέμα των κεφαλοπόδων βεβαίως που εξαρτάται και από τις συζητήσεις που θα λάβουν χώρα στην ε, μεικτή αυτή επιτροπή. Ελπίζω να ήμουν αρκετά πληρής, να σας ενημερώσω με συγκεκριμένα στοιχεία, να δώσω απαντήσεις. Αυτό που είναι σαφές, λέω κλείνοντας ότι μια αναδιαπραγμάτευση κατά την άποψή μας δεν ε, είναι κάτι πιθανό. Αναδιαπραγμάτευση σημαίνει ότι ξεκινάμε εκ του μηδενός, δηλαδή ότι η αλία διακόπτεται με εξίσου αρνητικές συνέπειες για κάποια τμήματα του στόλου και χρειάζεται ένας με 1,5 χρόνο διαπραγματεύσεις με τη Μαυριτανία. Ας δώσουμε μια πιθανότητα ε, στο πρωτόκολλο το να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα ε, τα σκάφη. Συνεχίζουμε τη συζητήση με την Ορδενία για να βελτιώσουμε το πρωτόκολλο. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να προωθήσουμε τη δυναμική, να μην τη σταματήσουμε άνευ εναλλακτική ε, λύσεω. Αυτά και ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ. Υπήρξαν κάποιες αντιδράσει. όσο μιλούσατε. Βεβαίως η Κομισιόν μάλλον θα λάβει απάντηση στα όσα είπε, κυρίως από τον εισηγητή, γιατί αυτός θα έχει την τελευταία κουβέντα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Θα ήθελα πω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αν είχε κάνει καλή διαπραγμάτευση και αν είχε ακούσει τους ενδιαφερόμενους δεν θα βρισκόμαστε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση όπου δεν επιδέχεται αναδιαπραγμάτευση. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω όλους που έλαβαν το λόγο, γιατί κανένας δεν αμφισβήτησε την έκθεση. Υπήρξαν ε, κάποιες αποχρώσεις στα σχόλια. Ε, η κυρία Λόβιν και ο κύριος Ρωμέβα υπέβαλαν παρατηρήσεις που έλαβαν απάντηση από την ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε ότι δεν καταλαβαίνει γιατί παραπονιόμαστε, γιατί υπάρχουν ποσοστώσεις, ε, θα, αλλιευ... θα πολύ περισσότερα ψάρια από ό,τι παλιά. Άρα καταρρίφθηκε το δικό σου επιχείρημα. Μερικοί συνάδελφοι έδωσαν ιδιαίτερη, ιδιαίτερο βάρος και σημασία στη θέση της Μαυριτανίας, κάτι που σέβομαι. Αλλά γιατί δεν δίνεται αντίστοιχη βαρύτητα και σημασία και στη θέση του Ευρωπαϊκού Ελληνικού Στόλου, γιατί οι Μαυριτανοί ήταν αρνητικοί και κατηγορηματικοί. Αλλά και εμείς το ίδιο και οι Ευρωπαίοι το ίδιο. Κάποιος είπε ότι οι Μαυριτανοί ήταν σαφές ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα. Δεν τους αρέσει τελεία και παύλα. Δεν υπάρχει περιθώριο λιγμών. Μα το ίδιο ισχύει και για μας. Το ίδιο ισχύει και για τα επιχειρήματα του Ευρωπαϊκού Στόλου. Ούτε και μας μας αρέσει. Και όμω φαίνεται ότι θα συνεχίσουμε τι συζητήσει. Και όχι μόνο συνεχίζουμε τι συζητήσει, αλλά εφαρμόζεται και η συμφωνία που δεν θέλαμε. Δεν νομίζω ότι είναι πολλά τα επιχειρήματα. Αλλά δεν θα πρέπει να συγχαίουμε τα εμπορικά επιχειρήματα με τα επιχειρήματα τα αναπτυξιακά. Ή λέμε να μην ερχόμαστε σε σύγκρουση με τον τοπικό πληθυσμό. Μιλάμε για τελείως διαφορετικά πράγματα. Και αυτό θα το μπορούσαμε να το επιλύσουμε θαυμάσια. Βιωσιμότητα και να μην έρθουμε σε σύγκρουση με, την, με τον τοπικό πληθυσμό. Ε, τότε ας αφήσουμε την ελευτική συμφωνία, να δώσουμε απλώς τα 70 εκατομμύρια να δείτε τι χαρούμενο ήταν ο τοπικό πληθυσμό, Αλλά αυτό είναι παράλογο. Τέλο, για αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μα είπε και πάλι ότι τηρεί το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και σε αυτό αγκιστρώνεται με νύχια και με δόντια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μα το ψήφισμα αυτό ήταν ε, ακριβέ και είχε νόημα σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Το έχουμε πει επανειλημμένος ότι αυτή η έκθεση αυτό το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει πια μείνει, έχει καταστεί παροχημένο από τα νέα επιστημονικά πορίσματα ανταποκρινόταν στην κατάσταση του 2009. Είχαμε έκτοτε πολύ πρόσφατες εκθέσεις και μελέτες που δείχνουν ότι δεν ευσταθεί η διαπίστωση της ε, υπερεκμετάλλευσης. Έχει αλλάξει η κατάσταση του αποθέματος χταποδιού. Επίσης είπε η Επιτροπή ότι έλαβε υπόψη τα αιτήματα των Μαυριτανών. Μακάρι να είχε λάβει εξίσου υπόψη και τα αιτήματα των Ευρωπαίων ε, αλλιών. Γιατί αν ως ε, πρωταρχικό στοιχείο της αξίας της συμφωνίας είναι το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό μας το προβάλλει ως επίτευγμα, μα φυσικά εννοείται. Αυτό είναι ένα θέμα που είναι οριζόντιο για όλες τις συμφωνίες. Δεν είναι κάτι που τιμά ιδιαίτερα αυτή τη φορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι κάτι κοινό. Επίσης αναφέρθηκε ότι οι συνθήκες είναι ισότιμες για, όλες τις, ε, για όλους τους στόχους. Με ίσως γι' αυτό δεν πηγαίνει κανένας ε, αλληλευτικός στόλος, γιατί είναι απαράδεκτες για όλους οι συνθήκες. Τώρα, μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυξήθηκε η ποσόστοση των πελαγικών από 250.000 στις 300.000. 150.000 είχε ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με βάση ποιες εκθέσεις. Αν τώρα μας το προβάλλει ως επίτευγμα ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 300.000 είναι κατά της βιωσιμότητας. Παλιά έλεγε πολύ λιγότερο. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι το σωστό. Ξεχάσετε τη βιωσιμότητα για να μας πουλήσετε ακριβώς το επιχείρημα ότι είναι σημαντικό ε, που αυξήθηκε η ποσότητα 300.000. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σκέφτηκε νωρίτερα ότι θα έπρεπε να έχει κάνει ένα σχέδιο διαχείρισης που να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των ειδών αυτών. Και τώρα, για τα κεφαλόποδα. Πολύ περίεργη κατάσταση. Περάσαμε από μία θέση που ήταν αυτή τη Επιστημονική Επιτροπή, στην άλλη θέση ότι οι Μαυριτανοί το διεκδικούν αποκλειστικά για αυτού. Από το ένα άκρο στο άλλο. Τότε, γιατί σε ένα χρόνο θα α, ε, κάνουμε νέα διαπραγμάτευση. Ή είναι μηδέν γιατί το θέλουν οι Μαυριτανοί, ή δεν είναι μηδέν. Το να είναι μηδέν και υπάρχει δυνατότητα αναθεώρηση δεν έχει νόημα και το σκέφτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα, θα μας στοιχήσει αυτή η αναδιαπραγμάτευση ή μήπως περιλαμβάνεται στα 70 εκατομμύρια αυτή η αναδιαπραγμάτευση του μηδενικού τάκ για τα κεφαλόποδα. Σε ό,τι αφορά την αλία θαλασσινών, σε τι μελέτε στηριχθήκατε. Γιατί λέτε ότι είναι πολύ πιο δύσκολα και ε, επώδυνα και τα πανηρά τα μέτρα για τα θαλασσινά. Και συνεχίζετε παρόλα αυτά. Για, τα, για το μερλούκιο, 4.000 τόνοι, για 11 σκάφη. Και δύο σκάφη μόνο καλύπτουν αυτή την ποσόστοση. Τι κατανομή θα γίνει μεταξύ των 11. Απο... Αποκλείται με 4 μόνο χιλιάδες τόνους μερλούκιο να ε, εξυπηρετηθούν 11 σκάφη. Επίση, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το πρωταρχικό είναι να μπορεί κανεί να λιεύει. Όχι, μα εδώ ήδη οι αλληλεί δήλωσαν ότι δεν του ενδιαφέρει να πάνε εκεί να ψαρέψουν. Είπατε ότι είναι δύο μόνο τα παραγαδιάρικα. Μερικοί έχουν, εμπορική, έχουν αλληλευτική άδεια, δεν δηλαδή θέλουν καν να ψαρέψουν. Επίση, λέτε ότι ένα τμήμα του πρωτοκόλου θα επηρεάσει αυτού που έχουν αλληλευτικό συμφέρον και άλλου όχι. Ένα τρίτο του, στόχου μας, του στόλου μα, είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι δεν είναι καθόλου βιώσιμη αυτή η κατάσταση και πολύ πανίρω μόνο για ένα τρίτο του στόλου. Δηλαδή 14 σκάφη που ουσιαστικά αλλιεύουν από τα 123. Δεν σα φαίνεται ότι παρά είναι ακριβό το τίμημα. Δεν σας φαίνεται υπερβολικό και ακριβό να πληρώνουμε 70 εκατομμύρια σύν την εισφορά του κλάδου μόνο για 14 από τα 123 σκάφη. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ συμφέρουσα αυτή η λύση. Επίσης, τι έγινε με τα 70 εκατομμύρια, τα πληρώσατε ή όχι. Και αν ναι, τότε γιατί αυτή η σπουδή όταν υπήρχε τρίμηνη προθεσμία για να βουλώσετε το στόμα ή ίσως ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να αποφύγετε το όχι του. Και ολοκληρώνω με μια ερώτηση που νομίζω ότι συνοψίζει τη συζήτηση και θα ήθελα μια απάντηση που μάλλον δεν θα είναι εύκολο να δοθεί. Δεν διαρωτήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν μια τόσο καταπληκτική συμφωνία, αν είναι τόσο καταπληκτική η συμφωνία, γιατί αρνούνται να πάνε να ψαρέψουν οι αλλοί. Αφού είναι τόσο καλή συμφωνία, τόσο θαυμάσια, γιατί δεν πάνε να ψαρέψουν οι αλλοί. Και μόνο αυτό θα έπρεπε να προβληματίσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα καταλάβει ότι δεν είναι τόσο καλή συμφωνία όσο νομίζει, είναι κακή και θα, έπρεπε να είχαμε αποφύγει αυτές τις δαπάνες εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν ήταν αναπτυξιακή βοήθεια θα έβγαζα πρώτο στο καπέλο μου. Αλλά δεν μπορούμε να δίνουμε αναπτυξιακή βοήθεια υπό το πρόσχημα μιας ε, συμφωνίας που είναι αμυγός ελευθερική, εμπορική. Ευχαριστώ. Ωραία. Άρα κλείνουμε αυτή τη συζήτηση. Προθεσμία για τροπολογίε είναι 29 Ιανουαρίου το μεσημέρι. Ψήφο στην Επιτροπή 18 ή 19 Φεβρουαρίου. Ψηφοφορία στην Ολομέλεια μάλλον το Μάρτιο. Κλείνουμε λοιπόν αυτό το σημείο. Και αφήνω το μικρόφωνο και πάλι στον πρόεδρο. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Ας περάσουμε στο επόμενο σημείο. Όπως διαπιστώνετε κι εσείς και είχα προβλέψει κι εγώ στην αρχή, έχουμε μείνει πίσω στο χρόνο. Οπότε το σημείο 7 της της διάταξης, την έκθεση Νικολέσκου, δεν θα προλάβουμε να τη συζητήσουμε σήμερα. Την αφήνουμε για αύριο που θα περάσει μετά το σημείο 12. Δηλαδή θα είναι το τελευταίο σημείο της αυριανής πρωινής μας συνεδρίασης στο σημείο 7. Οπότε μας έχουν απομείνει δύο ακόμη εκθέσεις που θα προσπαθήσουμε να τις διεκπαιρεώσουμε με ταχύτητα αστροαπή. Σημείο 5. Τροποποίηση του κανονισμού 812 για θέσπιση μέτρων σχετικά με παρεμπίπτοντα αλλιεύματα κήτο ειδών κατά την αλλία και για την τροποποίηση του κανονισμού 88 του 98. Ήδη ακούσαμε την παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Οκτώβριο. Τον Νοέμβριο έγινε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την έκθεση και σήμερα θα εξετάσουμε το σχέδιο έκθεσης του κυρίου Ρωμέβα Ιρουέδα, στον οποίο δίνω και το λόγο. Παρακαλώ, λίγη ησυχία. Αν θέλει κανείς να μιλήσει με την Επιτροπή, παρακαλώ εκτός εθούσης. Ευχαριστώ όλους όσους ε, είστε εδώ για την παρουσία σας και ευχαριστώ και όσους φύγουν για την απουσία τους. Θα είναι πολύ σύντομη συζήτηση πραγματικά. Γιατί μετά την πρώτη ανταλλαγή απόψεων και μετά από τις εκτενείς διαβουλεύσεις και με εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με την νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να δούμε με μεγαλύτερες λεπτομέρειες στους όρους της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τελικά καταλήγω στην απλούστατη πρόταση ότι θεωρούμε πως γενικά η πρόταση της ε, Επιτροπής είναι λογική σε ό,τι αφορά την προσαρμογή των διατάξεων στο νέο πλαίσιο της συνθήκης της Λισαβόνας. Οπότε, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθούν οι κατεξουδότηση πράξη για την προσαρμογή των προϋποθέσεων και των τεχνικών μέτρων για τη χρήση των ακουστικών συσκευών αποτροπής και επίση εκτελεστικών πράξεων όσον αφορά τη διαδικασία και τη μορφή υποβολή των εκθέσεων, στι οποίε υποχρεούνται να υποβάλλουν τα κράτη-μέλη. Και για να προσθέσουμε και εμείς κάτι, να συνεισφέρουμε στην ε, έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποβάλαμε δύο μικρούλες τροπολογίες που μπορούν, να θέλουν, να τις σχολιάσουν οι συνάδελφοι. Η πρώτη είναι τεχνική, η δεύτερη ίσως είναι πιο ουσιαστική και αφορά την... τον περιορισμό της εκχώρησης εξουσιών στην τριετία και όχι σε απεριόριστο χρονικό διάστημα. Και επίσης έχουμε την ενημέρωση, την τακτική. Αυτά. Είχαμε εκτενή συζήτηση και διαβουλεύση, παραλαμβάνω, με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το θέμα είναι πια όριμο για απόφαση, αλλά αν υπάρχουν σχόλια από τους συναδέλφους είμαι στη διάθεσή τους και περιμένω τα σχόλιά τους. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Αρσένης έχει το λόγο. ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Ρωμαίβα για την ε, δουλειά του. Έχω βέβαια μια παρατήρηση για την ε, ε, περίοδο της ισχύω των κατεξοδότησης πράξεων, που είναι τρία χρόνια. Το έχουμε ξανασυζητήσει νομίζω το θέμα αυτό και είχαμε πει ότι θα υπάρξει τροποποίηση των ε, τεχνικών προδιαγραφών ε, για τις συγκεκριμένες συσκευές ε, και νομίζω ότι η κατεξιότητες πράξη θα πρέπει να περιορίζονται στα τρία χρόνια, αλλά ίσως σε τούτη εδώ να είναι ειδική περίπτωση και θα ήθελα να το ξαναδούμε το θέμα αυτό. Παρόλα αυτά έχουμε... 10.000 κήτη που πεθαίνουν στην, ε, στα ευρωπαϊκά ύδατα. Ε, το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα αυτό και σε πλαίσια βέβαια τούτης της ε, έκθεσης, αλλά πάλι δεν βρίσκουμε λύση για τούτη τη μεγάλη απειλή. Υπάρχει και η έκθεση ISIS του 2010 που λέει ότι δεν υπάρχουν προϋποθέσεις από την σχετική οδηγία. Ε, μιλά μόνο για συγκεκριμένες ζώνες, κυρίως δηλαδή για τη Μεσόγειο. Υπάρχει πολύ, περιορισμένος, ε, πολύ περιορισμένη υποπτία και όπου γίνεται δεν γίνεται σωστά, γίνεται, με, γίνεται λάθασμένη ελεία, με λάθος τρόπο και βασίζεται α, πάρα πολύ στους δείκτες για τα παραλιεύματα. Κάποια κρατημέλη έδειξαν ότι αυτό δεν είναι επαρκές ως μέτρο ούτε αποτελεσματικό. Υπάρχει βέβαια και μια θετική αναφορά, μιλά για την ευαλτική και για τα αποτελέσματα εκεί που είναι αρκετά επικοδομητικά. Θεωρώ όμως ότι θα πρέπει να υπάρξει μια παρόμοια πράξη όπως αυτή η Ευρωπαϊκή Πράξη για την προστασία των θηλαστικών. Και στα πλαίσια αυτής της λισαβονοποίησης της συμφωνίας θα πρέπει να ζητήσουμε λοιπόν από την Κομισιόν να πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία και θα υποβάλω και κάποιες τροπολογίες ως προς αυτό. Η κυρία Φράγα έχει το λόγο. Ευχαριστούμε τον κύριο Αρσένη. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, τον κύριο Ρωμέβα, και να πω ότι η έκθεση είναι καλή, σωστή, δεν έχει πρόβλημα. Και για να μην, ξαναβαρώ, να, να μην ξαναλάβω το λόγο σε επόμενες συμφωνίες ε, για την, επιτρο... για την προσαρμογή στην επιτροπολογία, εγώ συμφωνώ με την τριετία. Δεν θέλω το δικαίωμα εκχώρησης ε, εξουσιών να είναι απεριόριστο. Θα πρέπει να υπάρχει ένα χρονικό όριο και αυτό το σχόλιο ισχύει για όλες ε, τις εκθέσεις ε, που θα έχουν ως αντικείμενο την επιτροπή στην επιτροπολογία, την, συγγνώμη, την προσαρμογή στην επιτροπολογία. Κύριε Αρσένη, τα άρθρα 90 και 91 είναι αυτά που διέπουν αυτή την περίπτωση. Οπότε είναι μια απλή περίπτωση προσαρμογής στην επιτροπολογία. Και αυτό ισχύει για όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις. Δεν πρόκειται για τίποτα ιδιαίτερο. Άλλος κανείς? Η Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και για την έκθεση που παρουσίασε ο κύριος Κατανοούμε τις ανησυχίες, κατανοούμε και την ε, ε, ανάγκη να υπάρξει συγκεκριμένη περίοδος ε, ισχύω των κατεξόδων συμπράξεων. Θα το δούμε βεβαίως πολύ προσεκτικά το θέμα αυτό. Για τα σχόλια τώρα που έκανε ο κύριος Ασένης, ο συνάδελφος την προηγούμενη φορά είχε πει ότι ίσως αυτά τα θέματα θα μπορούσαν να συζητηθούν όταν υπάρξει ανάκληση του ε, κανονισμού ε, προς το παρόν, μετά την μεταρρύθμιση. Προς το παρόν θέλουμε να πούμε ότι αυτό είναι αρκετά τεχνικό εγχείρημα σε ό,τι αφορά την, ε, τις ε, που έχουμε από τη συνθήκη της Λισαβόνας, οπότε δεν θέλουμε να ανοίξει περαιτέρω η συζήτηση πέραν δηλαδή των ε, κατεξουδότηση και των εκτελεστικών πράξεων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Συμφωνώ απόλυτα με τις προτάσεις του κυρίου Αρσένη και συμφωνώ με την ανάγκη να σημειώσουμε πρόοδο, όπως πρότεινε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να το αφήσουμε αυτό για την επιτροπολογία και να κάνουμε ένα νέο σχέδιο που θα συμπεριλάβουμε τέτοιου είδους μέτρα. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δεν είμαι καθόλου κατά της ουσίας. Απλώς στην περίπτωση αυτή καλύτερα να περιοριστούμε στο θέμα της επιτροπολογίας. Τώρα, για την τριετία. Θέλουμε να είμαστε συνεπείς και με τις άλλες αποφάσεις που έχουμε λάβει για την επιτροπολογία. Δεν υπάρχουν κάποια θέματα συνεκτικά. Γι' αυτό και χάρη συνέπειας προτείναμε την τριετία. Αυτό και αν έχετε να καταθέσετε τροπολογίες θα τις εξετάσω. Ούτε και εγώ πάντως βλέπω ιδιαίτερη δυσκολία στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ρομέβα. Στις 29 Ιανουαρίου το μεσημέρι, 29 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι, λίγη προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Αυτά με το 5 και περνάμε στο 6 τροποποίηση του κανονισμού 2187 του 2005 για τη διατήρηση των ελευθερικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων στα είδατα της Βαλτικής θάλασσας, των Belts και του Sound. Σήμερα θα ακούσουμε μια παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόταση τροποποίηση του κανονισμού. Ο κύριος Γεψένα ε, ή η κυρία, δεν ξέρω, είναι εκπρόσωπος που θα μας κάνει την παρουσίαση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Διακεκριμένοι Ευρωβουλευτές θέλουμε να σας παρουσιάσουμε την πρόταση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου όσον αφορά τη διατήρηση των ευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας στη Βαλτική, στα Bells και το Sound και μέσω και της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ενώσεως πρόσφατα ετοιμάσαμε τέτοια πρόταση στη γενική προσπάθεια που καταβάλλεται ευθυγράμμισης της νομοθεσίας που ισχύει με τη Συνθήκη για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Οι εξουσίες που έχουν ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο δυνάμει του κανονισμού αξιολογήθηκαν και αναταξονομήθηκαν σε μέτρα κατεξιζώτησης πράξεων και εφαρμοστικά μέτρα. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιορισμένη είναι, αφορά την ευθυγράμμιση του κανονισμού με τα προαναφερθέντα και θεωρούμε ότι αδίποτε τροποποίηση εκτός του πεδίου εφαρμογής της ε, ευθυγράμμισης θα πρέπει να παραμείνει στα πλαίσια ουσιαστικής αναθεώρησης τεχνικών ε, μέτρων μετά την αναθεώρηση ΚΑΠ. Βασικές αλλαγές της είναι οι εξής αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω εφαρμοστικής πράξης τη συμμόρφωση των εθνικών μέτρων με τους όρους που τίθενται στον κανονισμό. Οι διατάξεις που παρέχουν γενική εξουσιοδότηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσαρμόσει τους λεπτομερείς κανόνες για όλο τον κανονισμό άνευ καθορισμού του πεδίου εφαρμογή είναι κάτι που διαγράφεται. Η ανάθεση για τροποποίηση του παρατήματος 1 που αφορά τον ορισμό των γεωγραφικών περιοχών αφαιρείται σαν αναφορά, θεωρείται σαν κάτι περιττό, διότι οι γεωγραφικές περιοχές αυτές παραμένουν αμετάβλητες. Εξού και έλλειψη ανάγκης τροποποίησης του παρατήματος 1 και η τροποποίηση του προσαρτήματος 1 και 2 άνευ ε, τεχνικών προδιαγραφών από το παράτημα 2 πάνω στις κατεξισοδότησης πράξης. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και περιμένουμε πώς και πώς την καρποφόρα συνεργασία μεταξύ μας. Ευχαριστώ. Θέλει κανείς το λόγο για το θέμα. Ο κύριος Γκρουμπάρτσικ. Ευχαριστώ κύριε Πραδρέμα. Δική μου είναι η έκθεση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την σωστή της ε, προσέγγιση ό,τι αφορά την προσαρμογή ε, και διατήρηση των ελευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων στα ύδατα της Βαλτικής ε, θάλασσας, των Μπέλς και του Σάουντ. Και νομίζω ότι η βασική ιδέα, η κύρια ιδέα της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σωστή. Βέβαια, στο συγκεκριμένο κανονισμό τον 2187 του 2005 υπάρχουν κάποιες απειρχιωμένες διατάξεις που καλό θα ήταν να, να τις εξετάσουμε. Δεν μπορούμε να τις αφήσουμε. Θα πρέπει να τις τροποποιήσουμε. Αφορούν το άρθρο 14, εκεί που μιλάει για τις, για τις διαστάσεις των ψαριών. Εκεί έχουμε σαφή αναφορά των απορρίψεων και μέχρι στιγμής εφαρμόζουμε συγκεκριμένη πολιτική για τις απορρίψεις. Και αν ε, διαβάσουμε το άρθρο, λέει ότι δεν επιτρέπεται να, να παραμένουν στο, κατάθρο, στο κατάστρωμα ψάρια που δεν πληρούν τις διαστάσεις, αλλά θα πρέπει να, τις, να τα ρίχνουμε. Επαναλαμβάνω, τέτοιες απορρίψεις για, τα, για τη Βαλτική θάλασσα είναι καταστροφικές και απαράδεκτες. Και είχαμε πει ότι μέχρι το 2014 θα επιλύσουμε το πρόβλημα των απορρίψεων στην Βαλτική. Και υπάρχει και δεύτερη διάταξη που επιβεβαιώνει την πρώτη, ότι ε, τα μικρότερα ψάρια που δεν πληρούν τις διαστάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την παραγωγή ηχθιαλεύρων και δεν μπορούν να διατεθούν προς πώληση στις ηχθιαγορές. Αυτό είναι ακόμη πιο παροχημένη διάταξη και θα πρέπει αμέσως να αλλάξει. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε τη διατήρηση τέτοιων απερχιαμένων διατάξεων στον κανονισμό αυτό. Ένα άλλο θέμα είναι τα ανεξέλεγκτα αλλιεύματα, τα βιομηχανικά. Θα πρέπει να γίνονται οι σωστοί έλεγχοι τέτοιων αλλιευμάτων και το τελευταίο άρθρο που είναι το άρθρο υπερθυμών 28, που λέει ότι μέχρι την 1η Ιουνίου του 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διεξάγει ε, επιστημονικές μελέτες για τα δίκτυα και την επιρροή τους στην, ε, στα κοπάδια φαλενών. Από ό,τι ξέρω δεν έγιναν μελέτες σχετικές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε ε, θα πρέπει να διευρύνουμε και προς αυτή την κατεύθυνση την την έκθεση. Συγγνώμη κύριε Γκρουμπάρτζικ, ε, ξέχασα ότι ήσασταν εσείς ο συγητής και παρολίγο να μην σας δώσω το λόγο. Ο κύριος Κούν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πολύ σύντομα για τις παρατηρήσεις που έκανε ο κύριος Γκρουμπάρτσικ. Θα πρέπει να δούμε γενικώ το σύστημα της αλλαγής των τεχνικών μαέτρων. Και θα πρέπει να δούμε και σε σχέση με τη Λισαβόνα τι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή κατεξουδότηση πράξη ή εκτελεστικέ. Και βεβαίω πρέπει να έχουμε υπόψη μα και την κοινή ελευτική πολιτική. Τι γίνεται, περνάει, δεν ακούγεται η διερμηνία μου, να συνεχίσω. Υπήρχε ένα πρόβλημα με την αγγλική διερμηνία, αλλά εντάξει, τώρα λύθηκε. Συνεχίστε κύριε Κρίνου. Ένα πρώτο βήμα λοιπόν θα είναι να συμφωνηθεί στο Κοινοβούλιο ο βασικός κανονισμός, έτσι ώστε να είναι σαφές το τι θα γίνει, να δούμε τι θα γίνει και με τις ε, εκφορτώσεις, τι θα γίνει με τις απορρίψεις, με τα TFC, με την μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Όλα τα τεχνικά μέτρα θα πρέπει να τα δούμε ανά ε, περιοχή αλίευσης. Και αυτό βεβαίω θα είναι αρκετά μεγάλη δουλειά που μα περιμένει. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να πούμε τώρα ποιε θα είναι οι περιοχέ που μπορούμε ίσω να διαγράψουμε ε, αν θέλουμε να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ. Θέλει άλλο κανεί το λόγο. Ωραία, ευχαριστώ. Ολοκληρώνουμε αυτό το θέμα. Και ολοκληρώνουμε και την απογευματινή μας συνεδρίαση, γιατί όπως σας είπα το σημείο 7 θα το εξετάσουμε αύριο στην πρωινή συνεδρίαση. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τους διερμηνείς και αύριο, αν θέλει ο Θεός, λέει ο Πρόεδρος. Καλό σας απόγευμα.